Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο νωρί σήμερα το πρωί για αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Καθίστε παρακαλώ, ώστε να αρχίσουμε χωρίς να σπαταλάμε το χρόνο μας. Είναι 8.30. Ναι, το ξέρω. Ευχαριστώ που ήρθατε για την Επιτροπή μας. Λοιπόν, κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης για σήμερα. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα. Συμφωνούμε με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν σχόλια. Ωραία, ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν. Επόμενο σημείο. Έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας για το 2019. Όπως βλέπετε, η μόνη αλλαγή στο σχέδιο αυτό, το νέο, είναι ότι αφαίρεσα τις Παρασκευές. Πιστεύω ότι μπορούμε να οργανωθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας τις υπόλοιπες μέρες και αν χρειαστεί κάποια έκτακτη συνεδρία θα την προσθέσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε εδώ τις Παρασκευές. Συμφωνείτε? Εγκρίνεται αυτό το χρονοδιάγραμμα λοιπόν? Καλώς. Τώρα για το δεύτερο ήμιση του 2019. Δεν είναι μεν στα χαρτιά μας, στους φακέλους σας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στην επόμενη επιτροπή, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογέ, το Μάιο. η νέα επιτροπή θα συστηθεί κλπ. Οπότε εδώ πέρα εμεί μόνο για το πρώτο εξάμεινο αποφασίζουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεκτό. Καλώ. Ωραία. Βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος θα εργαστούμε. Ε, ιδιαίτερες ανακοινώσεις δεν έχω. Ίσως την επόμενη συνεδρίασή μας τον Οκτώβριο. Και τώρα Πάμε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα των εργασιών μας που είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπή μας σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και κοινοτομίας Ορίζων Ευρώπη. Είναι ένα από τα νομοθετικά προγράμματα που συνδέεται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η ΙΤΡΕ είναι η αρμόδια επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Εμείς συντάξαμε γνωμοδότηση. Ο κύριος Φανίστεροι είναι ο εισηγητή μας για τη γνωμοδότηση αυτή. Παρακαλώ κύριε Φανίστερο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, τόσο νωρί. Τι να κάνουμε, αλλά θα ξεκινήσω θετικά. Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που έχουμε τους φακέλους μπροστά μας. Ε, χρόνια τώρα δεν είχαμε τα χαρτιά αυτά μπροστά μας. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά, ρωτάει ο εισηγητής. Ναι. Ναι, προβλέπετε. Λοιπόν, δεν πρόκειται για τίποτα επαναστατικό, έτσι, αλλά πρόκειται για μια εξέλιξη. Πώς μαζί θα προχωρήσουμε με την περιφερειακή μας πολιτική, πώς θα συμπεριλαμβάνουμε τις περιφέρειες, τις πόλεις, σε όλες τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ένα σωρό προγράμματα. Το Horizon Ευρώπη είναι ένα από αυτά. Horizon 2020 ε, ήταν ε, πριν, τώρα έχουμε το Horizon Ευρώπη. Και είναι καλό που η Ευρώπη μπορεί να συνεργάζεται με περιφέρεις είχαμε την ε, συζήτηση και παλιότερα για το finishing touch όσον αφορά τις επιπτώσεις της περιφερειακής πολιτικής και ποιος είναι, ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει αυτή να πάρει τώρα. Είναι πολύ ωραίο να έχει κανείς το χρόνο στις διακοπές, το καλοκαίρι για παράδειγμα και να κοιτάξει τι έγινε εγώ να διάβασα αυτό, αυτή την έκθεση. Όσον αφορά την αξιολόγηση του προγράμματος Horizon 2020 και τις προτάσεις για τη νέα περίοδο. Εντάξει, δεν είναι κάτι που αναφέρει λεπτομέρειες για την κάθε περιφέρεια και την κάθε πόλη, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο ανάγνωσμα. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε τι γίνεται με συνεργασίες και πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόσθετη αξία της περιφέρειας όσον αφορά την καινοτομία, τη γνώση, τη θεμελιώδη γνώση, την εφερμοσμένη επίσης γνώση και πώς όλα αυτά καταλήγουν σε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Όντως τα πράγματα ε, βελτιώθηκαν την τελευταία περίοδο. Και είναι μια αναγνώριση. Δεν λέμε προσοχή για την περιφερειακή διάσταση, Έτσι κι αλλιώς ε, το Horizon 2020 θέτει πολύ καλές βάσεις. Με όλους τους εταίρους μας ε, στις περιφέρειες, στα διάφορα οικοσυστήματα τα ευρωπαϊκά κοινοτομίας βασιζόμαστε ώστε να αναπτύξουμε τις κατάλληλες πολιτικές για τις περιφέρειες. Είναι κάτι που βοηθάει και την επιχειρηματικότητα, τη γνώση, τη βιωσιμότητα, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής κλπ. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο. Είναι πολύ καλό λοιπόν να διαβάσει κανείς αυτή την έκθεση. Για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την περιφερειακή διάσταση. Αυτό είναι το κλαστικό για τη δικιά μας την Επιτροπή. Αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε, να υπάρχει αυτή η περιφερειακή διάσταση, η εδαφική διάσταση στην ομοθεσία, στο κείμενο το οποίο έχει συντάξει ο αρμόδιος εισηγητής. Τώρα, κατά τη γνώμη μας, η Ήτρε στο κείμενό της πρέπει αυτή την περιφερειακή διάσταση να την κατανείμει σε ολόκληρη την επικράτεια. Γιατί μιλάμε συνέχεια για την αριστεία. Αριστεία, αριστεία. Ωραία, πολύ καλό στο Horizon Europe, αλλά το 90% των χρημάτων στις χώρες μέλη πάνε ακριβώς εκεί. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, φοιτητέ από την Βουλγαρία. Μετά από πέντε χρόνια σπουδών. Τι θα κάνουνε τελικά θα φύγουν από τη Βουλγαρία. Δηλαδή θα μείνουν εκεί που έχουν πάει για σπουδέ, αν έχουν πάει έξω. Και έτσι υπάρχει διαρροή κεφάλαιο. Χάνεται η γνώση από τι χώρε. Και εφόσον ζούμε σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό με μεγάλα επίπεδα ειδίκευση, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανισορροπία στην Ευρώπη όσον αφορά τη γνώση, την ειδίκευση κτλ. Πρέπει η γνώση να κατανέμεται παντού, να υπάρχει στήριξη όλων των ε, προγραμμάτων, να έχουμε υπόψη μας την αριστεία, αλλά όχι μόνο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θέλουμε τους καλύτερους ερευνητές, αλλά γι' αυτό πρέπει να πληρώνονται. Τι άλλο βλέπω. Βλέπω ότι στο ορίζον Ευρώπη, πέρα από το όραμα και την αριστεία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την καινοτομία, που είναι το τρίτο σημαντικό σκέλος εντάξει, η έρευνα, αριστεία, ναι, να τα διευκολύνουμε όλα αυτά με χρήματα από την Ευρώπη. Μετά υπάρχει η καινοτομία, υπάρχει το Συμβούλιο Καινοτομίας. Αλλά αυτό πρέπει να φροντίσουμε να δραστηριοποιείται και στις περιφέρειες και τις πόλεις που μας ενδιαφέρουν εμάς. Και η γνώση έτσι οδηγεί στη συνέχεια σε παραγωγή, σε διάδοση και εφόσον ξεκινάει από την περιφέρεια είναι και πιο εύκολο αυτό να γίνει. Υπάρχει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο ακριβώς πρέπει να κοιτάει τι γίνεται στις περιφέρειες και τις πόλεις. Στην έκθεση αυτή λοιπόν προσπάθησα, στη δικιά μου την γνωμοδότηση μάλλον, να βάλω την περιφερειακή διάσταση. Τι μπορούμε να πετύχουμε με τα κονδύλια μας στο ορίζον Ευρώπη, αλλά και πώς αυτά τα κονδύλια μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα ταμεία, το κοινωνικό ταμείο για παράδειγμα. Με την Ήτρε και με τον εισηγητή και με τον εισηγητή για το δικό μας Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης μπορούμε να συζητήσουμε Με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επίσης πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μέσα από το μηχανισμό ορίζων Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά πρέπει και οι χώρες μέλη από μόνες τους να φροντίσουν για αποτελέσματα και, και αυτό πρέπει να διατυπωθεί στον κανονισμό που σύντομα θα επεξεργαστούμε και εμείς εδώ. Λέω και πάλι ότι οι προπτικές είναι πολλές και οι ανάγκες είναι πολλές η διάσταση της συνοχής πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ. Πολύ σημαντική αυτή η πρόταση για την απασχόληση και την ανάπτυξη, προκειμένου η Ευρώπη να έχει αποτελέσματα. Το Ταμείο Συνοχής επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη των λιγότερων ανεπτυγμένων περιοχών, στην Ανατολική Ευρώπη για παράδειγμα. Και ορίζουν βοηθάει όλες τις χώρες. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη ισορροπία, συμπληρωματικότητα. Θέλω να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη, τι πιστεύετε για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Οι σκιώδεις ηγητές. Η κυρία Ροντρίγκες είναι η πρώτη. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Λάμπερτ για τις αρχικές του προτάσεις που παρουσιάστηκαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο προπολογισμό της ε, Ένωσης. Νομίζω ότι ορίζον Ευρώπη είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, έχει καλά καθορισμένους στόχους αλλά θα ήθελα να εκφράσω και κάποιες ιδέες πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια στρατηγική ευρεία για σύγκληση σε όλη την Ευρώπη και να δώσουμε ευκαιρίες για αριστεία που να καλύπτονται όλοι. Να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να κατανείμουμε καλύτερα την υποστήριξη για δραστηριότητες στον τομέα της ερεύνας και της ανάπτυξης. Υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη και να αποφύγουμε μονομερείς ροές στην Ευρώπη από την περιφέρεια το κέντρο. Πρέπει να στηρίξουμε τον τέταρτο πυλώνα του προγράμματος Ορίζοντας για την Ευρώπη και να προσέξουμε ιδιαίτερα το ότι στην περίοδο εφαρμογής του προγράμματος τι θα γίνει, διότι στον ορίζοντα 2020 υπήρχε μεγάλη κίνηση, μεγάλη μετακίνηση και ο κόσμος προχωρούσε, μετακινείτο προς το βορρά της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε απλούστευση των συστημάτων, χωρίς να αγνοούμε τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε θέση να διασυνδέσουμε τους κανόνες εφαρμογής των διεθνωτικών ταμείων με τους μηχανισμούς συνοχής μαζί με τους κανόνες του προγράμματος ορίζοντας για την Ευρώπη. Να μειώσουμε το άχθος με αυτόν τον τρόπο, και να δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες για την χρήση ε, του ορίζοντα Ευρώπη και του Ταμείου του Αναπτυξιακού ε, για να βελτιώσουμε την επιστημονική ε, έρευνα και την απασχόληση του τομέα της έρευνας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και την έρευνα στον αεροδιαστημικό τομέα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Αεροδιαστημική Υπηρεσία να είναι αυτόνομη, να δούμε πώς μπορεί να χειριστούμε τους ωκεανούς και πώς οι απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να πραγματοποιούν έρευνα. Επίσης και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να υπάρχει θετική διάκριση. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ερευνητικό δίκτυο για αυτές τις περιοχές γιατί πολύ συχνά μένουν εκτός πλαισίων να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε έρευνα για τεχνολογία εχμής για να ενισχύσουμε την Ευρώπη και εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε συνεχείς επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες που να καλύπτονται όλοι και να παράσχουμε ευρή υποστηρίξη για διάφορες σχετικές στρατηγικές και τέλος θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτού του είδους οι επιστήμες δεν είναι λιγότερο επιστημονικές από τι άλλες επιστήμες που λέμε ότι είναι οι σκληρές ούτως είπε είναι επιστημονικές επιστήμες. Ε, συνάδελφε Κατάινεν, κυρία Κατάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την ε, πολύ επαγγελματική γνωμοδότηση που μας υπέβαλε. Πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος Καινοτομίας πρέπει να ισχυθεί και να έχει κεντρικό ρόλο για να υποστηρίζει τις επιστήμες. Ένας ρόλος πρέπει να αναγνωριστεί. Υποστηρίζω και τις προτάσεις του εισηγητού να κάνουμε τις δέουσες αλλαγές για να πετύχουμε το στόχο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ευθυγραμμίσουμε το εθνικό περιφερειακό επίπεδο για τα καινοτόμα συστήματα με το ευρωπαϊκό. Να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Χρειάζονται κατάλληλε συζητήσει πάνω σε αυτό. Δεν συμφωνώ απόλυτα όμω με τι ιδέε του εισηγητού όσον αφορά την υποστήριξη τη εδαφική ε, διάσταση. Όσον αφορά τα κριτήρια για αναθέσει, ε, συμφωνώ ότι δεν δημιουργείται εν κενό η επιστήμη και ότι η αριστεία στον τομέα της έρευνας χρειάζεται ε, και άλλη υποστήριξη στον επιστημονικό κόσμο. Όσον αφορά τα κριτήρια, πρέπει να είμαστε ακριβείς. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο πρόγραμμα Horizon. Και μόνο η αριστεία, η ποιότητα και τα αποτελέσματα είναι τα στοιχεία που πρέπει να αποτιμώνται και να έχουν σημασία. Η εδαφική ε, συνέπεια, το δαφι, ο εδαφικό αντίκτυπο είναι κάτι πρέπει να παίζει ρόλο και να λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση ενός προγράμματος. Και το εδαφικό αποτέλεσμα μπορεί να βελτιωθεί καλύτερα μέσω των μέσων και της ε, πολιτικής συνοχής προτείνει να συνεριβάλλουμε ανθρωπιστική καινοτομία και κοινωνική καινοτομία εντός αυτού του οικοσυστήματος και των σχετικών εργαλείων. Αυτή είναι πολύ καλή ιδέα για να προχωρήσουμε. Είναι εργαλεία κάτωθεν προερχόμενα που πρέπει να είναι ανοιχτά προς κάθε καινοτομία ανεξάρτητα από το τεχνολογικό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω και σας ευχαριστώ. Επόμενος και ηγητής που βλέπω έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχωνεύει το πρόγραμμα πλαίσιο και τους κανόνες για συμμετοχή σε μια ενιαία νομική πράξη και βελτιώνει και απλουστεύει την κατάσταση το ορίζον Ευρώπης θα ενισχύσει την επιστημονική τεχνολογική βάση της Ένωσης. Έτσι θα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα και θα πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη για τους σχετικούς στόχους. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της Ενώσης και τη βιομηχανία της και θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε θετικέ προτεραιότητες για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την υλοποίηση των πολιτικών της. Προσπαθούμε να διαθέσουμε τους κατάλληλους πόρους για τη συνοχή. Το Ευρώπη, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι ένα από τα προγράμματα. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα περίοδο χρηματοδότηση μεταφέρει πόρου από τον υπολογισμό τη συνοχή προ άλλα ταμεία και προγράμματα. Μέχρι 5% στο InvestEU και άλλα 5% από άλλα προγράμματα για τη μεταρρύθμιση που απαιτείται. 10 δισεκατομμύρια για το για το μέσο και για τη διασύνδεση τη Ευρώπη και για άλλα προγράμματα σχετίζονται με το πρόγραμμα Horizon. Έγιναν περικοπέ τη πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να παραμείνουν πάλι λοιπόν ποσά λοιπόν στην πολιτική συνοχή. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο προπολογισμό για τον ορίζοντα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Το Horizon Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει την αριστεία στην έρευνα και καινοτομία, ενώ η πολιτική συνοχή θα υποστηρίξει τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη διαδικασία τη καινοτομία, ούτω ώστε καινοτομία να διατεθεί στην αγορά τελικά, να διαδοθεί καινοτομία, η προσαρμογή τη καινοτομία κλπ. Όλα αυτά αναλάβουν χώρα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια συγκέντρωση των προγραμμάτων Horizon σε περισσότερε περιοχέ. Η πολιτική συνοχή που χρηματοδοτεί την έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να διωθεί ακόμα περισσότερο με στόχο την αύξηση τη δυνατότητα καινοτομία σε όλη την Ευρώπη και σε λιγότερε ανεπτυγμένε περιοχέ, όλο ιδιαίτερω. Υποστηρίζουμε ένθερμα αυτή την προσέγγιση και θα πρέπει πολιτική συνοχή να χρηματοδοτεί την αριστεία στι περισσότερο προχωρημένε, απομακρυσμένε περιοχέ και να μειωθούν οι διαφορέ μεταξύ περιοχών. Αλλιώ δεν θα πετύχουμε την κατάλληλη συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε Νταμάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το πρόγραμμα για την καινοτομία και την έρευνα θα πρέπει να κάνει πρωταγωνιστές τις πόλεις και τις περιοχές και τους πολίτες είναι κάτι απαραίτητο για βιώσιμη ανάπτυξη, για την απασχόληση, κυρίω για την ευημερία των πολιτών. Δεν θα υπάρξει κανένα σχεδιασμός που δεν λαμβάνει υπόψη ε, τη συνοχή, όπως βλέπετε, τις συνθήκες. Λοιπόν, όσον αφορά τη γνωμοδότηση, εγώ θα ήθελα να συμβάλλω βασιζόμενοι σε αυτά που έχουν πει, έχουν πει οι σκιώδεις στην Ήτρε. Και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εστίαση στην περιφερειακή και τοπική πτυχή θα ήθελα να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στους στόχους σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα να πετύχουμε τους στόχους των μηδέν εκπομπών αερίων μέχρι το 2050 και θα πρέπει κατηγορικά να αποκληθεί κάθε είδους χρηματοδότηση που υποστηρίζει λοιπόν τα ορυκτά κάψιμα. Ε, δεύτερον, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει ένα θεμελιώδη ρόλο στη βιομηχανία και στην αγορά που σίγουρα είναι σημαντικό αυτό αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από τις ανάγκες της κοινωνικές και από την αξία που έχει η ίδια η έρευνα. Λοιπόν, θα ήθελα να υπάρξει καλύτερη εξισορρόπηση του κειμένου, δίνοντας τις σωστές προτεραιότητες και θετώντα ένα μητρό που καλύτερα αντι... αντιστοιχεί ε, στις αξίες που συμπεριλαμβάνουν τις συνθήκες της Ένωσης. Από την άποψη της οικονομικής υποστήριξης και αυτή τη φορά θα ζητήσω να υπάρξει μια αναφορά αυτολεξή, ούτως ώστε να αποφευχθούν κερδοσκοπικές και τυχαίες επιχειρήσεις με τους διαθέσιμους πόρους ε, χρησιμοποιώντα χρηματοστικά μέσα που διατίθενται. Τελικά απευθύνω μια έκκληση να πρέπει ξανά να θέσουμε και εντό αυτού και το εργαλείο για τις μονοξέ επιχειρήσεις που είχε καλή επιτυχία. Θα... Φαίνεται ότι τώρα σαν να θέλουμε να το λησμονήσουμε. Πρέπει να έχει προτεραιότητα αν το υπογραμμίσουμε, μπορεί οι μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν στην πρόσβαση στου πόρου για την έρευνα και την καινοτομία. Δηλαδή, ρητά να αναφέρεται και να μην υπάρχει αμφισημία. Αυτά ουσιαστικά έχω να πω σαν παρατηρήσει και θα υποβάλω σχετικά ε, τροπολογίε για να συμβάλλω στι προσπάθειε που καταβάλουν ε, οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η Σκιώδη. Αλλά και η κυρία Μπρέσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι έλαβε υπόψη του, θεωρώ ακριβέστατα, τις ανάγκες που υπάρχουν να διασυνδέσουμε το μελλοντικό πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη με τις περιφερειακές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής Πιστεύω όσο πιο πολύ μπορούμε να συγκεράσουμε τα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτά που διατίθεται, τόσο το καλύτερο που απαιτήχουμε αποτελέσματα που ίσως θα μπορούσαμε να αυτή την πτυχή να την σάγουμε μέσω τροπολογίες για πραγματική διάδοση της καινοτομίας σε όλες τις περιοχές. Αποφεύγοντας λοιπόν την συγκέντρωση σε λίγες περιοχές, σε περιοχές που είναι ισχυρές και πρέπει να υποστηριχθούν διότι είναι οι πρωταθλητές μας στον κόσμο αλλά αν θέλουμε να γίνουμε πιο πρωταθλητέ, καλύτεροι πρωταθλητέ στον κόσμο από ό,τι είμαστε σήμερα χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα καινοτομία που διαδεθεί, θα διαδοθεί σε όλη την επικράτεια. Πρέπει να συνεργαστούμε. Θα πρέπει περιφερειακές πολιτικέ να κινηθούν προ την κατεύθυνση τη καινοτομία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν αν αυτή τη ενία είναι σημαντική η πρόταση των περιφερειακών οικοσυστημάτων και που θα μπορούσαν ε, θα μπορούσαν να είναι στιγμή που οι περιφέρειες και θα μπορέσουν να έχουν μια στρατηγική δική τους και να αποφύγουν να σπαταλούν τους πόρους σε πολλούς στόχους και μπορούμε έτσι να συγκλίνουν οι διάφορες πολιτικές. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε στο Στρασβούργο θα εγκριθεί το ψήφισμα που ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα θεματολόγιο, ένα πρόγραμμα για την Ήπεθρο, για τις περιφερειακές ζώνες και για τις ορεινές περιοχές. Όπως ήδη υπενθυμίστηκε από τη συνάδελφό μας, εάν θέλουμε να αναπτυχθεί η καινοτομία και σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ιδιαιτερότητα με την οποία κοινοί στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν αλλάζουν ανάλογα με τις περιοχές. Από τις αστικές περιοχές, εκεί που μπορεί να βοηθήσει το θεματολόγιο το αστικό να αναπτυχθούν καλύτερα τα προγράμματα για αυτές τις περιοχές, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τις περιοχές που είναι πιο αεροκατοικημένες, όπου εκεί η καινοτομία δύσκολα ε, ριζώνει. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούν να ανανεώσουμε τους πληθυσμούς, να αυξήσουμε τον πληθυσμό τους. Να δημιουργήσουμε πυρήνες αναπτυξιακούς και ανατομίας και στην Ήπεθρο. Όπως τα FEE χωριά, Smart Villages, που ο συνάδελφος Μπόγκοβιτς ε, ανέφερε και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σαγάγουμε μία τροπολογία που θα υπενθυμίζει αυτή ότι και με κοινού στόχους θα πρέπει να καθορίσουμε προγράμματα που μπορούν να προσαρμοστούν με τις ιδιαιτερότητες για την ανάπτυξη καινοτομία και έρευνα σε περιοχέ που έχουν φυσικά προβλήματα, που είναι απομακρυσμένες απομακρυσμένε περιφερειακά ή που είναι αεροκατοικημένε ε, και η ανάπτυξη εκεί είναι πιο παραδοσιακού τύπου. Με αυτόν τον τρόπο πραγματικά μπορούμε να έχουμε υπόψη να καλύψουμε όλε τι περιοχέ Ευρωπαϊκή Ενώσης και να δημιουργήσουμε την κατάλληλη κρίσιμη μάζα, ούτω ώστε να αναπτυχθεί η ε, καινοτόμα δυναμικότητα τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμενοι με τη σκιώδη Συγήτρια, θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε Εκτιμώντα πάρα πολύ τις προσπάθειες συναδελφού που ακολουθεί σίγουρα την ε, σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάλεπτη, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης και τους κοιόδης. Χαίρομαι που όλοι αναφέρατε και φυσικά και ο Λάμπερτ ότι στην Ένωση έχουμε αυτή τη φυγή εγκεφάλων από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης Και βεβαίως, βεβαίως, και εμεί το αναγνωρίζουμε. Οι ταλαντούχοι πάνε στην ε, Δυτική Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε. Πρέπει να στηρίξουμε όμως και το έρασμο ΣΥΝ. Και όλα αυτά βεβαίως. Αλλά όταν τα στηρίζουμε να μην ξεχνάμε και τη συνοχή. Γιατί αν ε, δώσουμε πολύ μεγάλη χρηματοδότηση στον ορίζοντα και δεν ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή, ούτω ώστε οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη διαφορά του, να αναπτυχθούν, θα αυξηθούν οι ανισότητε. Και άρα μια Ευρώπη διχασμένη. Πιο διχασμένη. Πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά. Και βεβαίω αυτό συνδέεται με την πολιτική για την έρευνα, την καινοτομία και την ε, ανάπτυξη. Στην Ένωση κάθε κράτος μέλος έχει, πρέπει να επενδύει σε αυτούς τους τρεις τομείς το 3% του ΑΕΠ του. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει. Και βεβαίω οι πιο ανεπτυγμένε χώρε ε, έχουν ήδη επιτύχει αυτό το στόχο. Αλλά οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε πόρο απέχουν. Στην Κροατία έχουμε 1,8 μόνο. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να στηρίξει αυτές τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να καταλήξουν σε αυτό το 3% επενδύσεων στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Και κατόπιν να υπάρξει μια αναρμόνιση μεταξύ αυτού του 3% και του ορίζον. Η συνοχή. Σε αυτή τη συγκυρία δεν πρέπει να χρηματοδοτήσει το ορίζον. Αλλά πρέπει να βοηθήσει τις χώρες ούτως ώστε να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ τους στην ε, έρευνα ανάπτυξη και και μετά να υπάρξει και εναρμόνιση. να δούμε πώς ο ορίζον θα βοηθήσει τις χώρες που μέσω του 3% στην ουσία χρηματοδοτούν περισσότερο τον ορίζοντα και να στηρίξουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες συμπληρωματικά, όχι μόνο μέσω της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανένα άλλο να θέλει το λόγο. Α, ξέχασα τον κύριο Όλμπριχτ. Ναι, κάτι άλλο που θέλω να ξέρω. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αυτό θέλω να σας πω. Θα υποβάλουμε σε ψηφοφορία την πρόταση να αυξηθούν οι πόροι για το νέο ορίζοντα. Από 80 σε 120 δις. Αλλά, όπως είπε η κυρία Μάλετιτς, ταυτόχρονα προτείνουμε οι πόροι για τη συνοχή να μείνουν στο ίδιο επίπεδο. Είναι λοιπόν μια συνολική λύση, ένα πακέτο. Ναι, μεν περισσότερα για τον ορίζοντα, αλλά πρέπει και ε, η πολιτική συνοχή να μείνει στο ίδιο επίπεδο. Γιατί όταν συζητάμε το θέμα αυτό πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. πρόεδρο. Βεβαίω σα ευχόμαστε να επιτύχετε, να περάσει αυτή η πρόταση. Ελπίζω να, να το επιτύχετε. Και ο κύριο Όπελ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, πολύ χρήσιμο αυτό το πρόγραμμα. Και πρέπει να συνεχίσει να ε, εφαρμόζεται εμποφελώς και στο μέλλον. Πρέπει να ενισχυθούν πολλές περιφέρειες. Να βοηθήσουμε τις ισχυρότερες να βοηθήσουμε και τις ε, πιο ε, αδύναμες να γίνουν και αυτές ισχυρέ. Διότι από ό,τι βλέπουμε, μόνο οι μεγαλύτερες χώρες, οι πιο ανεπτυγμένες αξιοποιούν αυτούς τους πόρους. Το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν ε, οι ανισότητες. Ορισμένες θα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες από άλλε θα υπάρχει φύγη εγκεφάλων, θα υπολείπονται. Εφόσον εμεί θέλουμε να έχουμε μια περιφερειακή πολιτική μέσω αυτού του προγράμματος, νομίζω ότι δεν επωφελείται επαρκώς και μάλιστα μειονεκτεί η περιφερειακή πολιτική από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Στηρίζω λοιπόν το συντάκτη γνωμοδότησης και πιστεύω ότι πρέπει να παράσχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη τι δυνατότητε να υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα και όλε τι περιφέρειες των κρατών μέλων. Πρέπει τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν όλε του τι περιφέρειες να συμμετάσχουν. Επίση. πρέπει να οριστούν ορισμένα κατόφλια ή συνολικά ποσά χρηματοδότηση για κάποιε περιφερειες κάποιες, ε, κάποια κράτη-μέλη. Και αν δεν μπορεί η συγκεκριμένη περιφέρεια, το συγκεκριμένο κράτος μέλος να αξιοποιήσει πλήρω αυτές τις ε, χρηματοδοτήσεις να μεταφέρονται <clears throat> σε άλλες περιφέρειες που έχουν καλύτερα προγράμματα. Γιατί αν το κάνουμε αυτό δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν θα διασφαλίσουμε τη χρήση περισσο... μεγαλύτερου ποσοστού των ε, διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ιστορία συμπεριλαμβάνεται και η γεωργία. δέκα δις επιπλέον για την ε, καινοτομία στον ε, τομέα της γεωργίας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σημαντικό όχι μόνο για τις πιο ανεπτυγμένες αλλά και τις λιγότερο χώρες. Πρέπει λοιπόν όλοι να τα ακούσουμε αυτά τα επιχειρήματα, να τα λάβουμε υπόψη και να καταλάβουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να αξιοποιήσουν τους πόρους του προγράμματος. Αυτό ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Howard. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στόχος του προγράμματος Horizon είναι να βοηθηθεί η έρευνα και η γνώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η εφαρμοσμένη έρευνα έχει παίξει μεγάλο ρόλο για την ε, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την κατασκευαστική βιομηχανία, ούτω ώστε να είμαστε πρώτο πόροι στην τεχνολογική έρευνα. Όμως, προειδοποιώ, οι άλλες ε, ανταγωνιστικές οικονομίες στον πλανήτη δίνουν πολύ περισσότερους πόρους για την έρευνα και για την αριστεία στην έρευνα από ό,τι κάνει σε αυτή την ε, συγκυρία έρευνα. Όπως είπε η κυρία Μάλετιτς, πρέπει να εμπλακούν και οι εθνικοί προπολογισμοί για την έρευνα, να συνδυαστούν, να δημιουργηθεί μια συνισταμένη όλων αυτών. Και πάλι όμως προειδοποιώ, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην εχμή των κατασκευαστικών κλάδων και της επιστήμης, θέλουν η έρευνα να γίνεται εκεί που είναι ε, οι κατάλληλοι επιστήμονε, οι κατάλληλοι ερευνητέ. Αυτό είναι ένα γεγονό, μπορεί να μας αρέσει, ένα γεγονό. Ο στόχος του προγράμματος Horizon σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική είναι να υπάρχει δυναμικό για αριστεία, δυνατότητα για αριστεία στις περιοχές που είναι στόχοι της ε, περιφερειακής. Αυτό πρέπει να είναι και όχι ε, να αντικαταστήσουμε την αριστεία με κάτι διαφορετικό δεν κερδίζουν οι διάφορες περιφέρειες και ούτε και η πρωτοπόρα επιστήμη κερδίζει. Πρέπει ο ορίζον να συνεχίσει να έχει αυτό το στόχο να βοηθάει την αριστεία. Πρέπει τα ερευνητικά ιδρύματα που είναι σε αυτό το επίπεδο, αυτά πρέπει να βοηθηθούν. Αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, στις περιφέρειες που υπάρχει ανάγκη. Σωστά υπόθηκε αυτό ούτω ώστε να μην χάνουν τους ταλαντούχους επιστήμονες. Δηλαδή, ποιο είναι το κόλπο. Να υπάρχει σωστό συνδυασμό τη περιφερειακή με την αναπτυξιακή πολιτική, με την πολιτική μας για την έρευνα και την αριστεία. Για να κερδίσουμε και σε δύο επίπεδα. Δεν είναι δυνατόν να αντιπαραθέσουμε αυτά τα δύο. Δεν θα λειτουργήσει. Γιατί τελικά Ορισμένα από αυτά τα ε, ερευνητικά ιδρύματα δεν έχουν απλώ ε, μια πεντηκονταετία πρωτοπορία, αλλά 800 χρόνια πρωτοπορία και κανεί δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαλόντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Λάμπερτ Φανίστελροϊ και τους Κιώδης. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Φανίστερο, γιατί εδώ και τόσα χρόνια έχει αφοσιωθεί σε αυτό το θέμα. Αυτές τις ε, συνεργασίες που μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ του προγράμματος πλαίσιο και των διαθροτικών ταμείων. Και χαίρεται ιδιαίτερα η Επιτροπή που προτείνονται τροπολογίες που πηγαίνουν ακόμη παραπέρα για να επιτύχουν επιπλέον αποτελέσματα από τον περαιτέρω συνδυασμό. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Φανίστελ Ρόι αναφέρθηκε στην ενδιάμεση ε, αξιολόγηση του Horizon 2020. Προέδρευσε αυτής της αξιολόγησης ο κύριος Λαμί και αναφέρθηκαν σαφώς οι ανάγκες περισσότερης συνεργασίας μεταξύ των ενωσιακών με τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα για να επιτύχουμε την μεγαλύτερη απόδοση, επίπτωση στην έρευνα και καινοτομία. Τις πολιτικέ συμπληρωματικέ δεν θα πρέπει να αντιπαρατίθενται. Πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και είναι στόχος μας αυτό και για το Horizon 2020 και για τις, προτήσεις, τις προτάσεις για τα διαθωτικά ταμεία αυτό το ξαναλέει το κείμενο για το ορίζον 20. Θέλουμε πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες, συνδυασμού που θα εισαχθούν για πρώτη φορά. Γι' αυτό μας χαροποιεί ότι ο εισηγητής σας έχει υποβάλει μια σειρά τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι τα κύρια σημεία γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος, αλλά μπορούμε να σας στείλουμε ή μάλλον να βάλουμε στο site μας επιπλέον σχόλια προς τις προτάσεις της ε, έκθεσής σας. Πρώτα απ' όλα η εδαφική διάσταση. Σε διάφορες τροπολογίες τονίζεται αυτό, αυτή η διάσταση. Εμείς ως Επιτροπή πρέπει να στηριχθούν τα βέλτιστα προγράμματα. Και αν το κάνουμε αυτό θα έχει επίπτωση στην ε, εδαφική διάσταση. Τα βασικά λοιπόν κριτήρια είναι τα κριτήρια αριστείας. Αλλά σε συγκεκριμένους τομείς, εφόσον θέλουμε να υπάρξει επίπτωση και μάλιστα ε, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένα εδάφη. Βεβαίω. θέλουμε να υπάρξει τέτοια επίπτωση. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι αυτά τα εδαφικά κριτήρια ένα γενικό κριτήριο. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ αριστεία από τη μία και εδαφικότητα από την άλλη. Αλλά όπου έχει έννοια και εμένα από αυτού, η περιφερειακή διάσταση βεβαίως είναι κάτι που θα λάβουμε υπόψη. Και αν χρειάζεται και σε ιδεολογικέ σκέψει αλλά και σε άλλα σημεία του προγράμματο πλαίσιο, για να είναι πιο σαφέ, <clears throat> στη διάθεσή σα. Να το βάλουμε. Θα το εξετάσουμε τουλάχιστον. Δεύτερον, προτείνουμε τη διευκρίνηση, συγκεκριμενοποίηση μια σειρά ορισμών. Βεβαίω, να εξετάσουμε την ε, τροποποίηση κάποιων ορισμών, γιατί κάποιοι κατά τη γνώμη μας ε, δεν έχουν ανάγκη περαιτέρω διευκρίνηση. Κοιτάξτε, όσο πιο λεπτομεριακοί γινόμαστε, τόσο περιορίζουμε την ε, ευελιξία κατά τη φάση εφαρμογής. Οπότε, το βασικό είναι να συμφωνήσουμε επί των στόχων. Και μετά θα δούμε πώς θα προσαρμόσουμε και τους ορισμούς στη νομική βάση. Και να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού υπερβολικές λεπτομέρειες για τους ορισμούς. Ωστόσο, εκεί που αναφέρεται το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας, δεν ξέρω τώρα αν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο σε έναν ορισμό, Θα μπορούσε όμως να μπει εκεί που μιλάμε στο πυλώνα 3 του Horizon 2020 ε, για το οικοσύστημα καινοτομία. Λέγεται έμεσα, ίσως δεν είναι αρκετά σαφές, για να επιτρέπονται οι συνεργασίες που προτείνει η έκθεση Φανίσταλ Ρόι. άλλος ε, τομέας, συμπληρωματικότητα, συμβατότητα, συνεργασίες μεταξύ του ορίζοντα Ευρώπη και τα διαθροτικά ταμεία επί των οποίων ξέρω τις προτάσεις που έχουν γίνει. Αναφέρθηκε ότι αυτές οι συνεργασίες δεν θα πρέπει να περιοριστούν μεταξύ του Κοινωνικού Ταμείου και του Horizon 2020 αλλά και σε άλλους τομείς μέσω του InvestEU και το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη όπου έχει έννοια να συνδυάζονται τα προγράμματα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, τροπολογιών του εισηγητή δίνουν πληροφορίες, διευκρινίζουν τι τύπου προγράμματα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό το συνδυασμό. Επί της ουσίας συμφωνούμε. Αλλά ίσως ε, να αποφύγουμε να δίδεται η εντύπωση ότι μόνο αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να μπορούν να συνδυαστούν με τον ορίζοντα Ευρώπη. Γιατί αναφέρεται το ERDF, το ESF και το EFRD. Και άλλα προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν δεν διαφωνούμε με την πρόταση. Αλλά πρέπει να καταστεί σαφέ ότι δεν θα είναι μόνο αυτά που θα συνδυάζονται, αλλά και άλλα. Φυσικά, καλοδεχούμενη είναι οποιαδήποτε διευκρίνηση. Όπως είπε και ο κύριος Φανίστελροε και οι διάφοροι σκιώδεις, καλωσορίζουμε κάθε προσπάθεια να εξαλειφθούν δυσχέρειες στην απόπειρα συνδυασμού προγραμμάτων που μπορεί να υπάρχουν στο υπάρχον πρόγραμμα πλαίσιο. Ως Επιτροπή θέλουμε να αξιοποιούνται όσο είναι δυνατόν οι δυνατότητες που προκύπτουν από την επικείμενη τροποποίηση του κανονισμού για τις κρατικές βοήθειες. Έτσι θα έχουμε περισσότερη συμβατότητα στο μέλλον. Επίσης, κάτι άλλο που υπάρχει και στην έκθεση. Η δυνατότητα μεταφορών πιστώσεων μεταξύ προγραμμάτων. Αυτό είναι μία δυνατότητα κοινή αξιοποίησης. Γιατί είπα ότι υπάρχει και η δυνατότητα όχι να γίνουν μεταφορές, να υπάρχει κάποια συνεργασία, δηλαδή ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτείται από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δηλαδή ένα πρόταση εγχειρήματο να ε, βοηθείτε από άλλο πρόγραμμα, όπως μέσω του προγράμματος ε, Σφραγίδα Αριστείας. Για παράδειγμα, θέλουμε στους εταιρικούς φορείς που δημιουργούμε να μπορούν να συμμετάσχουν και περιφερειακοί φορείς, κάτι που δεν ισχύει στο υπάρχον πρόγραμμα. Αλλά για τις μεταφορές πιστώσεων επανέρχομαι. Σημειώνουμε την πρόταση του εισηγητή, ιδιαίτερα για το άρθρο 9.8. Αλλά η μόνη μας ανησυχία είναι ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε ειδικά εγχειρήματα, γλυκές προτάσεις, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται σε ολόκληρα τα προγράμματα. Να μπορεί να μεταφέρεται ένα τμήμα του προπολογισμού ενός προγράμματος για να χρηματοδοτηθούν μια σειρά από project σε άλλο πρόγραμμα. Για να αποφύγουμε και κάποιες τεχνικές δυσχέρειες. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά διατακτικοί. Τέλος. Σημειώσαμε την πρόταση για την αλλαγή του προγράμματος, συγγνώμη, για την αλλαγή του πυλώνα 3. Το σημειώνουμε. Καταλαβαίνουμε την ε, επιχειρηματολογία. Κοιτάξτε, κάθε όνομα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Τώρα, μια που αναφέρθηκα στον πυλώνα 3, πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καινοτομία, Τον έφερε και ο κύριος Φανίστελροϊ, αλλά και άλλοι σκιώδεις. Προφανώς, συνεργασία με το Συμβούλιο αυτό πρέπει να υπάρχει. Αλλά για να έχουμε αυτή τη συνεργασία, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να είναι στον ίδιο πυλώνα, εντός του μπλοκ για το ε, οικοσύστημα καινοτομία. Έτσι θα προωθήσουμε την ευρωπαϊκή καινοτομία, το ευρωπαϊκό σύστημα καινοτομία, ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφερειών. Και ιδιαίτερα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, καινοτομίε τομεί, που είναι ακριβώς αρμοδιότητα του Συμβουλίου αυτού για την καινοτομία. Σε ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Στη διάθεσή σας ε, για να δώσουμε και περαιτέρω γραπτές διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φανίστερόη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Φτιάχνετε τη μέρα μου. Πράγματι, όντως πρέπει να βρούμε πώς θα έχουμε καλύτερη αξιοποίηση, πώς ε, θα επιστήσουμε την προσοχή στα θέματα που μας ενδιαφέρει. Τώρα, δεν μιλάμε για ανταγωνισμό, έτσι. Πόσα δηλαδή παίρνει ο ένας, πόσα παίρνει ο άλλος. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εντάξει, το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτά τα χρήματα. και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία ε, δεν λέω ότι θα πρέπει να κυκλοφορεί το χρήμα έτσι. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όσον αφορά τα χρήματα των φορολογούμενων και να προσπαθούμε με τα προγράμματά μας να τα αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Μιλάμε για συμπληρωματικότητα Τις τελευταίες δύο-τρεις περιόδους των ε, ταμείων είχαμε εξελίξεις. Άλλαξαν κατεύθυνση ή ενισχύθηκαν κάποιες. Και ήταν ανάγκη να γίνει αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν ε, η Ευρώπη να μένει πίσω στην ε, ανάπτυξη για την έρευνα. Και αυτά ακριβώ είναι που περιγράφονται και εδώ μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι. Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι πολλών ταχυτήτων και ακόμα λιγότερο Ευρώπη ε, πολλών ε, και διαφορετικών ευκαιριών. Διαφορετικών επιπέδων ευκαιριών δηλαδή. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Με την Ήτρε λοιπόν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε δυνατότητες για να πετύχουμε τους στόχους μας. Να παραμείνει η αριστεία, βεβαίως, είναι κεντρικό σημείο. Και το θέμα του ενστερνισμού επίσης παίζει ρόλο. Πρέπει κανείς να νιώθει υπεύθυνο. Αναφερθήκατε στο ψήφισμα. αν τροφοδοτείτε την έξυπνη δίκευση, έτσι τροφοδοτείτε και την οικονομία, έτσι τροφοδοτείτε και το κοινωνικό πυλώνα. Αυτά είναι λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε και να λάβουμε υπόψη μας αυτά που ζητάει και η περιφέρεια. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας που επίσης μπορεί να βοηθήσει τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν δυνατότητες λοιπόν πολλές. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πει ο, η Πρόεδρος πώς θα προχωρήσουμε ε, παραπέρα με το χρονοδιάγραμμα κτλ. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις. Ευχαρίστω. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 2 Οκτωβρίου. 6 ώρα το απόγευμα. Όχι Σαββατοκύριακο. Όχι Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να δουλέψετε το Σαββατοκύριακο. Ναι. Βλέπετε ότι ακόμα και το αναθερμένο χρονοδιάγραμμα της ε, Ήτρε δεν μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αν θέλουμε να μεταφραστούν τροπολίγου μας, ωραία, τι ώρα είπατε, στις 6 ώρα, δηλαδή μετά το τέλος των εργασιών, 6 ώρα το απόγευμα, 2 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα των εργασιών μας. Πρόκειται εξέταση της γνωμοδότησης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Ντόιτς από την Επιτροπή μας. Η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ντόιτς και ζητώ συγγνώμη που δεν υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Μπορείτε όμως να μιλήσετε ουγγρικά. Δεν ακούτε ουγγρικά, αλλά μπορείτε να μιλήσετε ουγγρικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν χρειάζεται να σας το παρουσιάσω. Νομίζω ότι το γνωρίζετε όλοι. Μιλάμε για έναν μηχανισμό πολύ βασικό γιατί βοηθάει ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους εξαιτία οικονομικών δυσκολιών, ε, τους βοηθάει να βρουν ξανά δουλειά, ενισχύει την κινητικότητα και ενισχύει επίσης και τις προσπάθειες που γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο από τις χώρες μέλη. Μιλάμε λοιπόν για ένα μέσο, ένα μηχανισμό που αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να νιώσουν το ωφέλη από το μηχανισμό αυτό στην καθημερινότητά τους. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα μηχανισμό ο οποίος βοηθάει να διορθωθεί ένα σοβαρό πρόβλημα, η ανεργία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάμε πολύ για την ανεργία. Πρόκειται όμως για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι στην Ευρώπη σήμερα. Συνεπώς, το να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς είναι ένα από τα κύρια καθήκοντά μας. Τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα έγγραφο, μια πρόταση κανονισμού δηλαδή, προκειμένου να συνεχίσουμε με το το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2020, γιατί πρόκειται για ένα έκτακτο ταμείο. Όλοι, νομίζω, συμφωνούμε με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρέπει να δούμε τώρα πώς θα απλοποιηθεί η εφαρμογή των κανόνων του Ταμείου αυτού. Με τη γνωμοδότησή μου ζητάω περισσότερη απλοποίηση, να συνεχιστεί δηλαδή αυτή η διαδικασία απλοποίησης. Ε, θα ήθελα το Ταμείο να συνεχίσει να χρησιμεύει και να βοηθήσουμε την διαδικασία νομοθετικής έγκρισης. Θα συνοψίσω σε τρία σημεία τα κεντρικά στοιχεία που έχουν να κάνουν και που συμπεριλαμβάνω στην γνωμοδότησή μου. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό να υπάρξει απλοποίηση των προϋποθέσεων πρόσβασης στα κονδύλια του Ταμείου αυτού. Συγκεκριμένα, Τώρα υπάρχει το των 250 απολύσεων που πρέπει να πέσει το νούμερο αυτό και να γίνει 150 απολύσεις. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές όταν χάνει κανείς τη δουλειά του αυτό συμβαίνει συνήθως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί οι απολύσεις δεν είναι μαζικές οπότε μία μικρομεσαία επιχείρηση δύσκολο θα απολύσει έτσι με μιας 250 άτομα. Γι' αυτό το όριο αυτό των απολύσεων θα πρέπει να περιοριστεί και αντί για 250 να γίνει 150. Πάντως θα μπορούσα να δεχτώ και μεγαλύτερη μείωση. Δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε μέτρα για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία και για να την επιταχύνουμε κιόλας. Στην πρόταση κανονισμού της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει Αναφέρει λοιπόν ότι η αξιολόγηση των ετοιμάτων σε συνάρτηση με την οικονομική συνεισφορά πρέπει να γίνεται as soon as possible, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η αλήθεια είναι πως αυτή η πρόταση είναι ιδιαίτερα σαφής. Όσο γίνεται πιο γρήγορα δεν σημαίνει τίποτα στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίρνει την απόφασή της σε 15 μέρες. 15 εργάσιμες μέρες, εντάξει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται καθυστερήσεις, μεταφράσεις κτλ. Οπότε τότε μπορεί να έχει 60 μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλύσει το αίτημα. Τώρα ισχύει αυτό. Λοιπόν, αντί για 60, εγώ προτείνω να βάλουμε 40 μέρες. Δηλαδή 15 συν 40, 55 μέρες. Σε 55 μέρες να υπάρχει απόφαση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι πιο αποδεκτό όταν υπάρχει μια κρίση, όταν κάποιος αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Καλό είναι να έχει γρήγορα και βοήθεια. Άλλη πρόταση που υποβάλλω έχει να κάνει με τη συγχρωηματοδότηση του Ταμείου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και το ποσοστό χρηματοδότησης θα πρέπει να παραμένει το 50% για τις χώρες εκείνες όπου υπάρχει αναρμόνιση μεταξύ των ε, ταμείων. Στη συνέχεια, θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο. Η σημερινή διαδικασία αρχίζει εφόσον έχει υπάρξει μαζική απόλυση. Εγώ όμως πιστεύω ότι υπάρχουν προδιαγραφές βέβαια που ορίζουν το τι είναι μια μαζική απόλυση, παρόλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την περίπτωση αυτή των 150 ε, απολύσεων και η διαδικασία θα πρέπει να ενεργοποιείται όχι μόνο εφόσον έχει ανακοινωθεί επίσημα, η απόλυση, αλλά από πιο νωρί ώστε να μπορέσει να γίνει η ένταξη των ε, απολυμένων σε κάποιο άλλο σχήμα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την ε, βοήθεια όλων και περιμένω και τα σχόλια των συναδέρφων για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που απολύονται να μπορούν όσο γίνεται πιο γρήγορα να ενσωματώνται και πάλι στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Το λόγο σου, Σκιώδης θα δώσω σύντομη, ένα τρίλεπτο έχετε στη διάθεσή σας γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα της ε, συνεδρίασής μας. Ο κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμπρότης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα της εργασίας του. Μας επιτρέπει να εξετάσουμε υπό άριστες συνθήκες το χαρτοφυλάκι αυτό, βλέποντας καταστροφικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρώπη τώρα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη από εργαλεία προσαρμογής αποτελεσματικά Εξ αυτού λοιπόν συνάγεται ότι ε, το εργαλείο αυτό είναι για την αντιμετώπιση των συνεπειών του, της παγκοσμιοποίησης είναι κάτι πολύ καλό και αποτελεσματικό ε, συνοδεύει τους εργαζομένους. Το επίπεδο επανένταξης των εργαζομένων που έχουν τύχη της υποστήριξης του μέσου αυτού είναι κάτι εξωσημείωτο. Ακόμα και στις περιοχές όπου η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή. Αυτό είναι αξιοσημείωτο ότι χρειάζεται επίσης ψυχολογική ε, υποστήριξη στην προσαρμογή των ανθρώπων, κυρίως ε, από αυτούς που έχουν ε, υποστεί τη συνέπειες θετικής αλλαγής των επιχειρήσεων. Λοιπόν, για την περίοδο 2020-2027 το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στο εργαλείο αυτό, ε, διευκολύνοντας τι διαδικασίε και του κανόνε. Το ίδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ελάφρυνση του τρόπου λειτουργία του εργαλείου και να διευρύνει την περίμετρο παρέμβαση. Έτσι μπορούμε να σημειώσουμε με μέγιστη ικανοποίηση ότι υπάρχει βούληση να μειωθεί, όπω είπε ο σε 250 τον αριθμό των απολύσεων που επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να προσφύγει στην υποστήριξη του μέσου αυτού. Εξάλλου, ε, σαν βουλευτής των υπερακτίων ε, επικρατιών, ευχαριστώ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπερπεριφερειακών περιοχών ε, ούσα άκρος ευέλικτη για το θέμα αυτό της δυνατότητας παρέμβασης. Δεχόμεθα θετικότατα τη συμπερίληψη των νέων καταστάσεων των ε, της ψηφιακής αλλαγής και της αλλαγής του κλίματος στο, στα πλαίσια αυτά. Έτσι η Ευρώπη θα μπορεί με καλύτερο τρόπο να προβλέψει τις συνέπειες που έχουν αυτά τα φαινόμενα. Έχω κάποιες προτάσεις ε, τροπολογιών για να συμπληρώσουμε το κείμενο. Κάποιες ε, τροπολογίες έχουν υποβληθεί από τη Μαρία Αλένα, Αλενά η οποία ε, εκπροσωπεί την Επιτροπή Απασχόλησης. Είμαστε πολύ εδώ που αναγνωρίζουμε ότι η ανεργία των νέων είναι και θα παραμείνει μεγάλο πρόβλημα. Θα προτείνω λοιπόν η βοήθεια του μέσου αυτού να ε, στηρίξει και τους άνεργους, ε, τους νέους που έχουν φύγει από το σχολείο και χρειάζεται υποστήριξη. Και σε εκείνους, που ε, είναι από περιοχές που είναι πάνω από 10% ενεργεία θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει και τους μισθωτούς των οποίων η θέση εργασίας ε, απειλείται από αναδιάθρωση της επιχείρησης. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο και ηγητής. Από το ECR έχουμε σκιώδη ηγητή. Όχι. Η κυρία Κατάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδιαμόρφωσε πράγματι ε, το μέσο αυτό για την αναπροσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση μείωση το όριο από 500 στους 250 απολυμμένους διεύρυνε και το πεδίο εφαρμογή του εργαλείου αυτού. Αυτό είναι θετικό, αλλά δημιουργείται ερωτηματικό ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ίσως πολλές πολλές μικρολεπτομέρειες θα αυξήσουν το διοικητικό άκθος και το κόστος που σχετίζεται με το πρόγραμμα και επίσης η διάρκεια επεξεργασίας ίσως να αυξηθεί. Έχει διευρύνει την κινητοποίηση και τη χρήση του Ταμείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό να μειωθεί το κατόφλιο περαιτέρω, όπως είπε ο εισηγητής, να πάμε από 250 απολυμμένους σε 150. Ε, θα ήθελα να ξέρω ποιες θα ήταν οι συνέπειες αυτής της αλλαγής στην πράξη και πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι και πώς θα στοχευθούν αυτοί οι πόροι. Είναι ένα ειδικό εργαλείο αυτό για ειδικέ περιστάσεις, το εργαλείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση για να μπορέσει να υπάρξει μια αντίδραση σε πολύ μεγάλες αναταραχές στην αγορά εργασίας. Εκεί μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση. κάτι κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν τα συστήματά τους για την αγορά εργασίας και για την εκπαίδευση παράλληλα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η επεξεργασία ε, των αιτήσεων, εξετάσεως των, εξετάσεων, των αιτήσεων συγγνώμη, πρέπει να επιταχυνθεί. Αυτή η επεξεργασία ε, τώρα διαρκεί μέχρι 6 μήνες. Αυτό δεν είναι ταχεία αντίδραση. Αυτά είναι τα σχόλια που έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βαλίνα δεν είναι εδώ. Η ε, κυρία Βάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα πολύ σύντομη. Είναι γνωστό ότι οι πράσινοι είναι πολύ θετικοί έναντι αυτού του ταμείου και συζητήσαμε με την συγκήτρια κυρία Ρένα και χαιρετίζω αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι <coughs> ότι πρέπει να διαβρεθεί το πεδίο εφαρμογή για να περάσουμε σε μια οικονομία αρνητικού, ε, χαμηλού άνθρακα και να δούμε και τις, να καλύψει και τις αρνητικές επιπτώσεις της, παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης, της και το γεγονός ότι καταβήκαμε στους 250 εργαζόμενους επίσης είναι θετικό, πολύ θετικό. Γιατί σε πολλές περιφέρειες δεν υπάρχουν τόσο πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε η κατάργηση ας πούμε 250 θέσεων εργασίας είναι ήδη μεγάλη ζημιά. Και χαιρετίζουμε και την έγκριση της αύξησης του προπολογισμού και την ε, ε, μείωση του χρόνου έγκρισης των προγραμμάτων που υποβάλλονται και όλα αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάτο. Η κυρία Μάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όπω γνωρίζουμε, ο στόχο ο γενικό του προγράμματο του Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση είναι να δείξουμε αλληλεγγύη και να παρασχεθεί υποστήριξη σε εκείνους που χάνουν την εργασία τους και στους αυ... αυτόνομους εργαζομένους που ε, μπορεί να πέσουν θύμα των αναδιαφθρώσεων. Είδαμε ότι οι εργαζόμενοι ότι στο, στο, στο πετσί τους νιώθηκαν τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, όπως τις αλλαγές των εμπορικών ροών στον κόσμο, η ε, οικονομική κρίση, η χρηματοπιστική κρίση και ότι αυτά έχουν αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση. Και όχι μόνο αυτό, σοβαρότατα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο προβληματισμού εντοπίζει το συνδυασμένο αποτέλεσμα τη παγκοσμιοποίηση που συνδέεται με το εμπόριο και με τι τεχνολογικέ αλλαγέ και ότι αυτοί είναι οι βασικοί κινητήρε, ε, ότι χρειάζονται εκπαιδευμένα χέρια και μείωση των θέσεων εργασίας που χρειάζονται λιγότερα προσόντα. Άρα χρειάζονται εργαλεία ενδεδειγμένα για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παράπλευρες αρνητικές συνέπειες που τοφοδοτούνται από πιο ταχεία αλλαγή ε, τεχνολογική. Σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας θα πρέπει να προβλέψουμε αυτές τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης και να βελτιώσουμε συνεπώς τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Λοιπόν, όσο έχει στον παρόν προγραμματισμό το μέσο ε, μπορούμε να βελτιώσουμε διάφορα σημεία. Θέλουμε αποτελεσματική υποστήριξη των εργαζομένων. Θα πρέπει να συμφιλιώσουμε, να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε του τιτογενού τομέα, όπου εκεί αντίκτυπο ενδεχομένων κρίσεων ε, έρχεται πιο καθυστερημένο σχέση με το βιομηχανικό τομέα. Για να δώσουμε επαρκή προστασία σε αυτού του εργαζομένου και στου αυτόνομου εργαζομένου, θα πρέπει να προβλέπονται μέτρα διαφορετικά προστασία. Θα πρέπει εκεί που χρειάζεται να υπάρχει μια διε... Ε, εκεί που βλέπουμε μεγαλύτερη διεύρυνση τη αγορά, ε, να αντιμετωπίζεται και η διαταραχή του τουγενή τομέα. Θα πρέπει και να ακολουθηθούν προληπτικά μέτρα. Θα πρέπει να επεκταθεί η επιλεξιμότητα για τα μέτρα υποστήριξης όλους τους εργαζομένους και αυτούς που έχουν ε, ορισμένου χρόνου και ορίστου χρόνου συμβάσεις ή και τους προσωρινούς εργαζομένους και τους αυτόνομους. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε ότι σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει το μέσο αυτό να υποστηρίζει την συνοδεία ή την κοινωνικο-οικονομική μεταλλαγή των διαφόρων περιοχών και ζωγραφικών ζωνών και διαφόρων τομέων επαγγελματικών που κυρίως πλήττονται όσον αφορά την απασχόληση. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία κινητοποίησεως Εξετά... θεωρήθηκε ότι είναι πολύ μακροσκελή και πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάφορα κάτι μέλη είπαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στην ε, εμβάθυνση τη ανάλυση των διαφορων περιοχων και ζωγραφικων ζωνων και διαφορων τομεων επαγγελματικων που κυριως πληττονται οσον αφορα την απασχοληση εν παση περιπτωσει η διαδικασια κινητοποιησης εξετα θεωρηθηκε οτι ειναι πολυ μακροσκελη και πλευρα τη ευρωπαικη επιτροπη διαφορα κατι μελη ειπαν οτι αντιμετωπισαν προβληματα στην εμβαθυνση τη αναλυση των περιστασεων που, δημιούργησε το, που δημιούργηκαν το πρόβλημα. Πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα οικονομική και, θα και θεσμική των αρμοδίων φορέων και θα πρέπει να, να διευκολυνθεί, ε, να χορηγείται η τεχνική βοήθεια πριν να υποβληθεί καν η αίτηση. Θα πρέπει να, κοινο, θα πρέπει να αντιδρούν αμέσω τα κράτη-μέλη, ώστε να υποβάλουν και ένα αίτημα χωρί να υπάρχει καμία καθυστέρηση. Το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Α, ο κύριος Φανίστελ, σύντομα παρακαλώ. Μα εγώ πάντα είμαι σύντομος. Καλή είναι η προσέγγιση του συναδέλφου. Αλλά, κοιτάξτε, αν ε, κατεβάσουμε το όριο στους 150, θα έχουμε τόσες αιτήσει. Μήπως θα πρέπει το ταμείο αυτό να συνδυαστεί γενικότερα με τις προσπάθειες καταπολέμησης της ανεργίας. Γιατί όλα μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Κοιτάξτε, στην ε, ε, Ολλανδία έχουμε βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις εργαζομένους στον τραπεζικό τομέα που πολύ σύντομα θα εκταμιευτούν και βλέπουμε ότι και η Air France έχει πάρει χρηματοδοτήσει γι' αυτό. Πρέπει να συνδυαστεί με την δράση του κοινωνικού ταμείου. Γιατί αυτά κάνει το κοινωνικό ταμείο. Βοηθάει τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και υπάρχουν δύο επίπεδα γιατί το κοινωνικό ταμείο είναι σε επίπεδο περιφερειών, ενώ, το ταμείο αυτό για την παγκοσμιοποίηση είναι σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε, αν το κατεβάσουμε στο 150 ε, θα έχουμε πάρα πολλές αιτήσει και θα πρέπει να εξετάσουμε ε, κάθε φορά θα λέμε γιατί την κάνουν αυτές τις απολύσεις. Είναι η παγκοσμιοποίηση ή είναι ότι η εταιρεία λειτουργεί καλύτερα και έχει περισσότερα κέρδη με, με λιγότερους εργαζόμενους λόγω της αυτοματοποίησης και της χρήσης της τεχνολογίας της τι θα κάνουμε λοιπόν. Αυτά είναι περισσότερα αυτά που κάνει το κοινωνικό ταμείο, αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη, ακόμη και οι περιφέρειες. Γιατί έχουν κάποια κοινωνική πολιτική. Τώρα είναι ένα ε, επι, επιμέρους όργανο που λειτουργεί αυτόνομα διαφορετικά. Κοιτάξτε, η προσπάθεια ε, να ε, καταρτιστούν οι εργαζόμενοι για να βρουν μια νέα δουλειά, άμα απολυθούν, είναι περισσότερο δουλειά του κοινωνικού ταμείου. Γιατί κοιτάξτε, έχουμε τόσο πολλέ απολύσει σε τόσο πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη 150 εργαζόμενων, που τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ε, ε, ε, μια σκέψη κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Οτσάνοβα από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση. Θα κάνω σχόλια στην πρόταση. Το κατόφλιο. Κάναμε πολλές ε, μελέτες για να δούμε ποιο πρέπει να είναι το όριο και εξετάσαμε την κατάσταση που είναι πολύ διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη και μειώσαμε στο μισό από 500 εργαζόμενους το κάναμε 250. Αυτό την κάνει πιο χρήσιμη για τα μικρά κράτη-μέλη, λιγότερο ε, ενδιαφέρουσα για τα μεγάλα κράτη-μέλη, γιατί δεν θα υπάρχουν επαρκή πόροι για όλους, αλλά σημειώνουμε αυτά που υπόθηκαν και όλες τις απόψεις. Η διάρκεια έγκρισης. Είναι πολύ τεχνικό. Ίσως μπορώ και κατηδίαν ε, να σας εξηγήσω. 15 εργάσιμες ε, στην ουσία είναι αδύνατο ε, μην ξεχνάμε ότι μόνο για τη μετάφραση όλες τις γλώσσες θέλουμε τρεις εβδομάδε. Μόνο για την μετάφραση. Λοιπόν, θα θέλαμε περισσότερο από αυτό που προτείνεται. Αλλά είναι πολύ τεχνικά αυτά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε κάτι δίαν. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας, δηλαδή για τη στήριξή σας, τις πρότασή μας, για τη σχηματοδότηση, για την ε, εναρμόνιση μεταξύ G.F και η ESF, γιατί ακούσαμε τις γνώμες των εμπλεκομένων και θεωρούμε ότι αν υπάρχει μια κοινή, κοινά ποσοστά χρηματοδότησης, είναι καλύτερα για την περίοδο μετά το 2020. Σημειώνω ότι κατά πλειοψηφία στηρίζεται την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή και τα αίτια που προτείνονται τώρα για την επιλεξιμότητα μίας αίτηση, ε, οικονομία χαμηλού άνθρακα, ψηφιοποίηση κτλ. Αλλά αποφασίσαμε να μην παραταθεί η χρήση του ταμείου μας για τους needs γιατί νομίζουμε ότι τώρα υπάρχουν ε, άλλες δυνατότητες, άλλα ταμεία, το ESF συν και άλλα προγράμματα που καλύτερα μπορούν να στοχεύσουν τους νέους αυτούς. Το οποίο, το οποίο ούτως ή άλλως οι διαστάσεις του ε, μειώνονται λόγω της ε, οικονομικής ανάπτυξης που έχει σημειωθεί. Υπήρξαν κάποια σχόλια και θέλω να κάνω δύο διευκρινήσεις για τον τραπεζικό τομέα που ανέφερε ο κύριος Φαν Λίστεροι και ε, αυτό που υπόθηκε για τη στήριξη εταιριών. Δώσαμε χρηματοδοτήσεις σε τραπεζικούς όχι λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά λόγω των υποπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης γιατί το Ταμείο μας αυτό ασχολείται με αυτές τις περιπτώσεις. Και οι Ολλανδοί που έκαναν αίτηση την αιτιολόγησαν ακριβώς ως επίπτωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τώρα είπατε ότι στηρίξαμε κάποιες εταιρείε. Το Ταμείο μας δεν στηρίζει εταιρείε, μόνο απολυμένους. όχι τις εταιρείε αυτές καθεαυτές. Πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Πρόκειται για εργαζόμενους, Ευρωπαίους εργαζόμενους, που εργάζονται εδώ στην Ευρώπη, που έχουν απολυθεί λόγω αρνητικών εξελίξεων. Στο μέλλον θα διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή, γιατί δεν υπάρχει κανένα ορισμό τη παγκοσμιοποίηση. Εμεί τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε κανένα ορισμό τη παγκοσμιοποίηση. Άρα στο μέλλον δεν θα καλύπτει μόνο περιπτώσεις επιπτώσεων παγκοσμιοποίησης. Νομίζουμε το ότι, ότι το ταμείο μας είναι ήδη πολύ γνωστό ιδιαίτερα από όσους έχουν ωφεληθεί από τις χρηματοδοτήσεις του. Γι' αυτό έχει πια ένα, ένα όνομα. Είναι γνωστό το όνομά του ως Ταμείο για την Προσαρμογή της Παγκοσμιοποίησης. Άρα επειδή όλοι το ξέρουν έτσι θα διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή γιατί θεωρούμε ότι όλα σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση τη σήμερα ημέρα. Ευχαριστώ κύριε Ντόιτς για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια, χωρίς να επεκταθώ ιδιαίτερα. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση αυτή. Εγώ προσωπικά σχολίασα κάτι και θα το επαναλάβω. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι συμπληρωματικό, οδρά συμπληρωματικά, προκειμένου να βοηθήσει, να βοηθήσει τη διαχείριση μιας αρνητικής κατάστασης. Να βοηθήσει την επανένταξη των απολυμένων στην αγορά εργασίας. Πρόκειται όμως και για το εξή. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και χρήματα από τις περιφέρειες, από τη συνοχή, για να δημιουργούνται νέες θέσει απασχόλησης. Συνεπώς υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης και μάλιστα πιο κατάλληλε για να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση και η απασχόληση συνολικά. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό μηχανισμό, επιμένω, και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία του. Τώρα ακούσαμε και πιστεύω ότι είναι θετικό ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη διάσταση των νέων, των νέων ανέργων. Τέλος, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, Πρέπει να δούμε τα τεχνικά ζητήματα περισσότερο. Ίσως κάποιες πτυχές να μην είναι σαφείς, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αιτήματα πρέπει να δοθεί συνέχεια. Όταν όμως οι μεταφράσεις είναι ήδη έτοιμες τώρα, έχουμε στη διάθεσή μας 60 μέρες για να ανταποκριθούμε. Και εδώ είναι που λέω ότι δεν πρέπει να λέει as soon as possible, όπως λέει το κείμενο τώρα, για να αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει συγκεκριμένη προθεσμία, που εγώ προτείνω να είναι 15 εργάσιμες μέρες για να πάρει την απόφασή της. Θα μπορούσε να ήταν και 20, ξέρω εγώ, και 17, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχει αυτό το ασαφές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πιέζει ο χρόνος, όπως πάντα. με τις γνωμοδοτήσεις μας. Οπότε, ε, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Απασχόλησης, προτείνουμε προθεσμία 3 Οκτωβρίου, 5 ώρα το απόγευμα, για την υποβολή τροπολογιών. Και παρακαλώ στα αγγλικά οι τροπολογίες σας, αν γίνεται, για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε έτοιμοι με την γνωμοδότησή μας πριν ψηφίσει η Επιτροπή Απασχόλησης. Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα είναι η προθεσμία. Ωραία. Ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση και συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η παρουσίαση της γνωμοδότησης, του σχεδίου γνωμοδότησης για την θέσπιση του προγράμματος Invest EU. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής είναι, είναι δύο. Είναι η Επιτροπή Προπολογισμών και η Οικονομική Επιτροπή που συνεργάζονται. Δικιά μας εισηγήτρια, συντάκτρια γνωμοδότησης, είναι η κυρία Κέστιν Βέστφαλ. Οπότε θα σας δώσω το λόγο σε εσά πρώτα απ' όλα, έτσι, για να κερδίζουμε χρόνο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας πω κάτι που είναι γνωστό, αλλά θέλω να το τονίσω από την αρχή. Τα διαφθορτικά ταμεία στόχο έχουν να βελτιώσουν τη ζωή των εργαζόμενων. Οι περιφέρειες δημιουργούν από τη μία θέση απασχόληση, βελτιώνουν τις υποδομές, καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή και στηρίζουν τα πανεπιστήμια, αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή μας αγωνίζεται ούτω ώστε να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα στήριξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων στο μέλλον, ακόμη και αν μειωθεί η χρηματοδότηση. Και από ό,τι φαίνεται, στο μέλλον θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε λιγότερα προγράμματα γιατί θα υπάρχουν λιγότεροι πόροι. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί προσπαθώ να εκφράζω, να εκφράσω ε, σοβαρέ ανησυχίε λόγω αυτού του πλαισίου για την πρόταση τη Κομισιόν για το InvestEU, η οποία πρόταση θέλει να μοχλεύσει ιδιωτικέ επενδύσεις μέσω εγγύσεων. Αυτό έχει έννοια. Σίγουρα βοηθάει τη χρηματοδότηση ορισμένων εγχειρημάτων. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα βοηθήσουν τους Δήμους και τις περιφέρειές μας και τις πόλεις μας να ε, βελτιώσουν την κατάσταση κατά τη γνώμη μου. Οι διαρθρωτικοί πόροι με την αποκεντρωμένη ε, διαχείρισή τους είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που προτείνει το Invest EU. Γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, απορρίπτω την ιδέα τα διαρθρωτικά ταμεία να αξιοποιηθούν για να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος Invest EU. Και συμφωνώ έτσι με τους δύο εισηγητές μας για το γενικό κανονισμό. Ναι στην ε, ιδέα να δημιουργηθούν συνδυασμοί, αλλά όχι στα σχέδια να μπλεχτούν αυτοί οι δύο ε, πηγές χρηματοδότησης. Γι' αυτό διαγράφω αυτό που λέγεται ε, τμήμα των κρατών μελών, Member State Compartment. Ο συντάκτη της Επιτροπής μας πρέπει να προστατεύσω τα δικά μας διευθυντικά ταμεία. Πολλές ιδέες του InvestEU μου φαίνονται καλές. Υπάρχουν ε, πολλές δυνατότητες βελτίωσης σε σχέση με το ΕΦΣΙ και το ΕΦΣΙ 2. Για παράδειγμα, θαυμάσια ιδέα να υπάρχει μια πλατφόρμα για ε, παροχή συμβουλών, advisory hub, να ε, δίνει συμβουλές για τα επενδυτικά προγράμματα. Καταλαβαίνω ότι όσοι ε, διαβάσουν αυτά που υπάρχουν σε αυτήν την πλατφόρμα θα διαβάσουν όχι μόνο τι δυνατότητε έχουν να λάβουν χρηματοδότηση από το InvestEU, θα μπορούσε Εάν κάποιος δεν μπορεί να ε, κάνει αίτηση για την InvestEU, θα μπορούσε να ζητήσει χρηματοδότηση από τα διεθνωτικά ταμεία. Εάν ε, θα βοηθούσε αυτή η πλατφόρμα τους ενδιαφερόμενους να στραφούν προς την κατάλληλη χρηματοδότηση, θα ήταν καλό. Καταλαβαίνω την... Ε, ότι η πρότασή μου, η οποία συμφωνεί και με τις προτάσεις των ε, κυρίων εισηγητών να αλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό τη δομή του InvestEU. Γι' αυτό η, η γνώμοδότησή μου εστιάζει ιδιαίτερα σε αυτά τα σημεία. Και ευχαριστώ την Πεάτα που έκανε καταπληκτική δουλειά επί των λεπτομεριών, κοίταξε παντού στο κείμενο, ούτως ώστε να αφαιρέσει παντού αυτά που αφορούσαν αυτό το τμήμα για το Member State Compartment και να τα διαγράψει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ γενικά τη γραμματεία. Ευχαριστώ ε, και τους συναδέλφους για τη βοήθεια που θα μου δώσουν στην περαιτέρω επεξεργασία αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές. Η κυρία Σπυράκη. Θέλει να μιλήσει κανείς εκ μέρους της κυρίας Σπυράκη. Όχι, σήμερα. Καλώς. Ο κ. Βανίστερ Συμφωνώ απόλυτα με τη γενική προσέγγιση. Πιθανότατα λοιπόν στο τέλος της περίοδου σχεδιασμού πρέπει να γίνει ανάλυση που δεν αποδίδουν ε, σωστά τα, τα κράτη-μέλη. Και ίσως έχουν τη δυνατότητα τα χρήματα που δεν έχουν ξοδέψει να τα βάλουν στο InvestEU. Το Horizon, Horizon Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό, διότι εκεί ο σχεδιασμός γίνεται στην αρχή. Ίσως συμφέρει κάποια κράτη-μέλη που δεν έχουν ξοδέψει τα ποσά, που είναι πολλά από αυτά, στα μισά της περίοδου να εξετάσουν την κατάσταση και να πούν. Κάποια δεδομένη στιγμή, στα μέσα της περίοδου, λέω εγώ, τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν μια ανάλυση και να πούν χρησιμοποιούμε το μέσο στο τέλος, στο τελευταίο χρόνο, να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Ερωτηματικό είναι, δεν έχω άποψη. Ίσως και αυτό μπορεί να συζητηθεί. Μπορεί να τεθεί αυτό σαν θέμα. Ευχαριστώ. Επόμενος κέρδης. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Κυρία Τόμασιτς, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόγραμμα Invest Europe θα δώσει κάποιες εγγυήσεις για να στηρίξει τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων βασίζεται σε εμπειρίες που αποκτήθηκαν με τα Ταμεία Εύση. Σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο μέσο πρέπει να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω μιας δομής που αναδιαρθρώνει και ομαδοποιεί και θέτει σε κοινό πλαίσιο τα εφιστάμενα μέσα. Η προτάση του κ. Βέστφαλτ σχετίζει τα δύο επενδυτικά μέσα και μου αρέσει αυτό και αναφέρεται και στο ρόλο των περιφερειών στο InvestEU. Συμπεριλαμβάνεται και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διαφόρων εφαρμοστικών ε, φορέων. Ξέρουμε από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μείωση των πόρων για όλα τα ταμεία ΕΦΣΥ κατά 10% εν συγκρίση με το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπεται ότι οι πόροι συνοχής από το ΕΦΣΥ μπορούν να διατεθούν για το Invest EU ή να μεταφερθούν σε άλλα ταμεία ή άλλα μέσα. 5% των συνολικών ποσών υποκοινή διαχείριση μπορεί να συμβάλλουν ε, στη χρηματοδότηση του Invest EU. Φοβούμαι ότι αυτό θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αποσύρουν τους πόρους από τα προγράμματα συνοχής. Μία απλή μεταφορά οδηγεί σε μείωση των πόρων ε, για προγράμματα συνοχής και αυτό δεν είναι λύση. Γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή να διαγραφεί το τμήμα των κρατών μελών όπως αποκαλείται από το InvestEU. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ εν συντομία θα ήθελα να συμμετάσχω στη συζήτηση. Έχω κάποιες σκέψεις να εκφράσω. Πρώτα απ' όλα Αυτός ο συνδυασμός των ταμείων ΕΦΣΥ και του ε, Invest Europe. Αυτό αναφέρεται στην πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ηγηθεί στην προσπάθεια και όχι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αναλάβει τους ε, σχετικούς κινδύνους και πώς θα μεταμορφωθεί σε ιονή τράπεζα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Αν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, να προωθήσουμε τις επενδύσεις, αυτό είναι κάτι που συνεπάγεται κάποιους κινδύνους και κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτούς τους κινδύνους στην περίπτωση του Ταμείου ΕΦΣΥ και αυτόν που έχει ε, πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το να το αναλάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ήταν καλή λύση. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Και ίσως να είναι κάπως πολιτικά ορθόδοξο αυτό που θα πω. Οι πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει προτεραιότητα στην Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, στις μεγάλες χώρες γενικά. Θα ήθελα να βρούμε έναν τρόπο, ούτω ώστε τα μικρότερα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες που θα προσφερθούν από αυτό το Ταμείο. Διότι είναι γεγονός ότι οι μικρότερες χώρες χρειάζονται πολύ περισσότερες επενδύσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ανεργίας, φυγής εγκεφάλων κλπ. Χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν την τελευταία διετία από την Κροατία. Και ο αριθμός των κατοίκων μας από 4,5 εκατομμύρια έχει πέσει στα 4 εκατομμύρια. Αυτή είναι δραματική μείωση. Άρα είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις. Χρειάζονται επενδύσεις κυρίως οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Το ΕΦΣΥ έχει απλουστεύσει κατά κάποιο τρόπο τις διάφορες διαδικασίες. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε μελλοντικές προτάσεις και προγράμματα και να μην λησμονούμε και τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες. Συχνά αναφέρεται ότι, θέλουμε, ε, ότι δεν θα επενδύσουμε σε υποδομές πλέον, αλλά είναι προφανές κάτι αναγκαίο αυτό, διότι και υποδομές οδηγούν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε μεγαλύτερα έσοδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες στη Μεσόγειο που αντιμετωπίζουν πολύ ψηλή ανεργία, κυρίως ανεργία των νέων και βασίζονται αυτές οι χώρες πολύ στον τουρισμό. Χρειαζόμαστε επενδύσεις σε αυτό τον τομέα και την κατάλληλη υποδομή που στηρίζει αυτό τον τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αν θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους στα νησιά της Ελλάδας, Φερρυπίν, ή ε, τον κόσμο στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Το καλοκαίρι επεσκέφθην την Νότια Γαλλία και είδα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τη χώρα αυτή στον τομέα τον τουριστικό. Ελπίζω να λάβετε υπόψη κάποιες από τις προτάσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Βέστφαλ, σας στηρίζουμε εκπεφρασμένα. Δεν είναι δυνατόν να μειώνονται οι πόροι των διαθροτικών ταμείων και να πηγαίνουν στο ΕΦΣΙ. Δεν είναι η πρώτη απόπειρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και κατά τη διαδικασία Omnibus ε, το απορρίψαμε. Η κυρία Κρέλ ε, ήταν παρούσα και δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να έχουμε τις ίδιες προτάσεις. Δηλαδή πάντα η περιφερειακή, η διαθροτική, η πολιτική συνοχή να αποδυναμώνονται και να δημιουργούνται νέα όργανα που είναι προσανατολισμένα προς την οικονομία της αγοράς. Είναι επίθεση κατά της πολιτικής συνοχής. Και πρέπει να το λέμε. Πρόκειται για όλα τα επιτεύγματα που ε, μέσω της πολιτικής ε, για τα διευθυντικά ταμεία. Όλα αυτά τα θέματα που έχουμε επιτύχει για το κοινωνικό τομέα, η αστική διάσταση, η περιβαλλοντική διάσταση, όλα τα επιτεύγματα που έχουμε εισαγάγει μέσω της εργασίας της Επιτροπής μας στα ταμεία καταργούνται. Αν δω πώς λειτουργεί το ΕΦΣΥ, πέρα από την ε, επανειλημμένη κριτική του ελεκτικού συνεδρίου, βλέπουμε ότι δεν γίνονται επαρκείς ε, κοινωνικές επενδύσεις για κοινωνικές ε, υποδομές. Δεν προκύπτουν μέσω του ΕΦΣΥ. Οπότε, θα μπορούσαμε να ήμασταν ιδιαίτερα επικριτικοί έναντι αυτών προτάσεων. Και θα εξετάσουμε τις προτάσεις αυτές και θα καταργήσουμε όλες τις προτάσεις που αφορούν μεταφορές πιστώσεων. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Νταμάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά, η ιδέα ενό προγράμματο επενδύσεων για τι εσωτερικέ πολιτικέ ένωση, σαν μόνο σύνολο κανόνων, πρέπει να επιστρέψει μια σαφή απλούστευση. Από την άλλη πλευρά, όπω και το ΕΦΣΙ, που παρουσίασε διάφορα προβλήματα και αυτό το παράγωγό του δεν είναι ε, άνευ αυτών. Παραμένουν πολλές σκιώδεις περιοχές όσον αφορά το πώς θα πρέπει να παρέμβουμε. Η διαφάνεια, η προσθετικότητα, ο σεβασμός αρχής συνοχής που βγαίνει από τις συνθήκες και ε, το αποτέλεσμα μόχλευσης θα πρέπει στεναρά να αντιδράσουμε για να μην τροφοδητηθούν κερδοσκοπικέ κινήσει που είναι επιζήμιε για την πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση του δημοσίου χρήματο για την υποστήριξη επιχειρήσεων χρηματοπιστωτικών πολύ παρακινδυνευμένων. Μετά υπάρχει ένα στοιχείο σημαντικό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν στι εγγυήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με ένα ποσοστό των δικών του πόρων. Ε, όπως είναι τα διαθετικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ε, λοιπόν, ε, και αυτά είναι χρήματα που χρησιμοποιούνται στη συνοχή. Προορίζονται σε περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες. Για την Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να συμμορφώνονται, ε, να, να αφήσουν το κάτω μέρος να κινηθεί και να βοηθήσει σε παρεμβάσεις όχι μόνο σε μονομενιχτούσες περιοχές, αλλά εκεί που υπάρχει, πρέπει να αποφύγουμε να γίνονται οι παρεμβάσει και υπάρχει μεγαλύτερο κέρδο αντί στι περιοχέ μειονεκτούσε. Θα πρέπει στο επίκεντρο τη συνοχή να είναι οι πραγματικές ανάγκες των μειονεκτουσών περιοχών και περιφερειών. Και κάτι άλλο που είναι απαράδεκτο και γι' αυτό θα υποβάλω και τροποποίηση είναι πιο συνολός του Κοινοβουλίου. Να θυμηθούμε ότι ο μόνος εκλεγμένος φορέας είναι το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αφήσει εκτός, μας έχει κάνει θεατέ, παθητικού θεατέ το Κοινοβούλιο. Θα θέλα να πω ότι με το InvestEU θα δημιουργηθεί μια κατάσταση που δίνει πολλές εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να μπορεί εκ των πραγμάτων να δράσει σαν τράπεζα. Αλλά αυτή δεν είναι η φύση της ούτε δική της αρμοδιότητα, αν θέλουμε να σεβαστούμε συνθήκες ενώσεως. Αυτή η, αυτή η ευθύνη που ανέλαβε μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της δίνει ιδιαίτερες ε, εξουσίες όπου ε, για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να επικυρώσουν οι επιτροπές, η ανάθεση των κινδύνων κλπ. είναι ευαίσθητα στοιχεία και πολύ σημαντικά στοιχεία ε, και χρειάζεται προσεκτική χρήση αυτών για τη χρήση του δημοσίου χρήματος και γι' αυτό θα υποβάλω τροπολογίες που με τρόπο καλύπτουν τις διάφορες πτυχές που ανέφερα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς. Τώρα έχω και εγώ τα δικά μου προσωπικά σχόλια, επιτρέψτε μου. Έχοντας ακούσει τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών, έχω μια ερώτηση προς την ε, συντάκτρια. Προσπαθούμε να πετύχουμε ε, συνεργασίες, ε, κοινή αξιοποίηση δράσεων επενδυτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά η επιλογή μεταφοράς κονδυλίων από τα διευθυντικά ταμεία στο Invest EU γίνεται σε θελοντική βάση. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένη καμία χώρα να το κάνει όντω. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες θα μπορούσαν όμως να χρησιμοποιήσουν και τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Εδώ σε αυτή την επιτροπή πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να σκεφτούμε το θέμα της ευελιξίας και των δυνατοτήτων που έχουν οι χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μέσα. Έχω στο μυαλό μου το γεγονός της κοινής αξιοποίησης ότι είναι μόνο σε εμβριακό στάδιο. Οπότε, η ερώτησή μου είναι, μπορούμε να την αφαιρέσουμε αυτή την πρόταση. Άκουσα τη θέση των σχεδόν εισηγητών ότι θα είναι απόφαση της Επιτροπής Ρέτζη. Όλα αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε με ευφύ τρόπο και να είμαστε σε θέση να σκεφτούμε επόμενα βήματα της πολιτικής συνοχής. Ο κύριος Όλμπριχτ έχει ζητήσει το λόγο επίσης και μετά κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ. Δεν έχω ερώτηση, πρέπει να πάω στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά κάτι άλλο. Έχω κάποιες προτάσεις για την συντάκτρια γνωμοδότησης. Κοιτάξτε, εγώ που ετοιμάζω το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει το ερώτημα να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι το InvestEU. Η συζήτηση έγινε και λέγαμε πρόκειται για ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για όλες τις πολιτικές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Είναι ένα πρόγραμμα εγγύησεων. Δεύτερον, τι γίνεται με τις πολιτικές από τις οποίες αφαιρούμε κονδυλιά. Όχι όπως στη συνοχή, αφαιρούμε χρήματα και δημιουργούμε παράθυρα στο ρίζον για παράδειγμα, για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις κτλ. Τότε πώς θα χειριστούμε αυτό το παράθυρο, πώς περιλαμβάνεται στον προπολογισμό, γιατί αφαιρείται από μια πολιτική και πηγαίνει σε μια άλλη πολιτική, που είναι στα χέρια άλλων, όχι της δικής μας γενικής διεύθυνσης. Οπότε είναι θέμα διαχείρισης και το άλλο που ρωτάμε εμεί οι Τι θα γίνει με την πολιτική συνοχή. Συζητήσαμε πάρα πολύ για τα χρηματοδοτικά μέσα μέσα στην πολιτική συνοχή. Υπάρχουν το Τζέσικα κτλ. Το ξέρουμε. Και ξέρουμε επίσης τι σημαίνει να βάλουμε κάποια χρήματα τα οποία θα μείνουν εκεί γιατί είναι δύσκολο να δαπανηθούν. Μερικές χώρες μέλη, και έχει δίκιο η Πρόεδρος, οι χώρες φοβούνται ότι θα χάσουν τα χρήματα Οπότε για αυτά είναι μια διέξοδος να αποταμιεύσουν χρήματα, να τα σώσουν. Δεν θέλω να επικρίνω το InvestEU. Απλώς θέλω να ζητήσω από τη συντάκτρια γνωμοδότησης να φροντίσει να μπει στην έκθεση από την Επιτροπή μας να υπάρξει ένα παράθυρο συνοχής. Γιατί σε θελοντική βάση θα πηγαίνουν τα χρήματα στο Infest EU χωρίς παράθυρο συνοχής. Οπότε θα πηγαίνουν σε κάποια άλλη πολιτική. Θα φεύγουν από την πολιτική συνοχής και θα πηγαίνουν σε μια άλλη πολιτική. Και αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να σκεφτούμε τα εθνικά κονδύλια και την πολιτική συνοχής. Να σκεφτούμε και να συζητήσουμε για τους μηχανισμούς. Τι δηλαδή επενδύσεις μπορούν να γίνουν καλύτερα μέσω τραπεζών και ποιε όχι, αλλά πάντα στα πλαίσια της συνοχής, ακόμα και αν υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός. Οπότε να μην φεύγουν τα χρήματα χωρίς να υπάρχει παράθυρο συνοχής στο Invest EU. Αν δεν υπάρχει παράθυρο, τα χάσαμε. Θα εξαφανίσονται από την πολιτική συνοχή στα κονδύλια αυτά και θα χάνονται. Πρέπει να φύγω γρήγορα, αλλά ήθελα να τα έχω πει αυτά στην ε, συντάκτρια γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε. Κυρία Κρέλ τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να συμμετάσχω στη συζήτηση, αλλά σχετίζεται με αυτό που κάνουμε στον γενικό κανονισμό. Εκεί βλέπουμε ότι θέλουμε να γίνουν αυτές οι διαγραφές. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες ότι ίσως κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν ότι θα χάσουν κάποιες ε, πιστώσεις. Αλλά αν τους δώσουμε ευθύ εξ αρχής τη δυνατότητα να αφαιρούν πόρους από το InvestEU και να το πάνε, α, ε, συγγνώμη, πόρους από τα διεθνωτικά ταμεία και να το πηγαίνουν στο InvestEU, τότε τα κράτη-μέλη θα αξιοποιήσουν αμέσω αυτή τη δυνατότητα. Γιατί είναι πολύ απλούστερε οι διαδικασίε του InvestEU. Όλε οι αρχέ, ε, όλοι οι πολιτικοί στόχοι τη Ένωση, κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, όλα αυτά θα τα παρακάψουν εντελώ. Στέλνοντα ε, του πόρου στο InvestEU και τότε μπορώ να πω αγαπητή Επιτροπή πάρτε 20% από τους πόρους της συνοχής δεν τα θέλουμε, κάντε ό,τι θέλετε δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή η αντιμετώπιση μας τι ρόλο παίζουμε τότε ούτως ή άλλως θα περικοπούν κατά 10% τα κράτη, οι πόροι για τη συνοχή τα κράτη-μέλη τουλάχιστον θα πρέπει να κάνουν την κάθε προσπάθεια για να αξιοποιήσουν τουλάχιστον αυτούς τους ε, μειωμένους πόρους Βεβαίω, βεβαίω. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Έρασμο, με τον InvestEU, με τον Ορίζοντα, με το Life. Βεβαίω, τα λέει αυτά. Τα λέει αυτά ο γενικό κανονισμό. Και έτσι διευκολύνεται και η χρηματοδότηση τη έρευνα που δεν θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν ε, για προγράμματα που δεν θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στον ορίζοντα. Αλλά βλέπω ότι διάφορα κράτη-μέλη λένε μα τα λίγα χρήματα που έχω για την περιφερειακή πολιτική τα χρειάζομαι για περιφερειακά προγράμματα και έχω αρκετές δυνατότητες ε, άλλες όπως η Τζέσικα και τα άλλα εντός της πολιτικής συνοχής για να τα αξιοποιήσω. Προεδοποιώ, υπάρχουν ε, πιέσεις από πλευράς ε, συγκεκριμένων κρατών μελών να καταλάβουμε ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε αρμόδιοι για περιφερειακή πολιτική για μια κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Λόγος ύπαρξής μας δεν είναι να ε, χρηματοδοτούν κάποια κράτη-μέλη τερατώδη προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική συνοχή. Οπωσδήποτε όταν θα συζητήσουμε το γενικό κανονισμό πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πρέπει η πολιτική συνοχή να παραμείνει όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη το λόγο ύπαρξής μας εδώ ως Επιτροπή. Προειδοποιώ. Αυτό το InvestEU να μην το υποτιμήσουμε. Και τι επιπτώσεις θα έχει για την πολιτική συνοχή η λειτουργία του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει και η πρόεδρος. Η κυρία Μάλετιτς. Μια φράση να πω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε και άλλους συνάδελφους, πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Πώς είναι τόσο περίπλοκη η πολιτική συνοχή σε συγκρίση με το InvestEU, εν συγκρίση με τον ορίζοντα. Τα κράτη-μέλη προτιμούν να δίνουν χρήματα στο InvestEU και το Horizon παρά να προσπαθούν να τα χρησιμοποιήσουν μέσω της πολιτικής συνοχής. Με το νέο CPR δεν βλέπω απλούστευση περιπλέκεται το σύστημα σε σχέση με τα προηγούμενα. Έχουμε περισσότερους όρους από τις, τις ε, παρούσες προοπτικές, δημοσιονομικές προοπτικές. Πρέπει να πλουστευτεί η πολιτική συνοχής. για να γίνεται σωστή κατανομή των πόρων από τα κράτη-μέλη. Ήταν μια φράση περί απλουστεύσεως, λέει η Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να πω κι εγώ κάτι, μια φράση. Και σχετίζεται με τις μελλοντικές συζητήσεις για τα διάφορα ταμεία και ε, το διάφορο... και τι κοινέ προβλέψει για το μηχανισμό κοινών προβλέψεων. Είχαμε κάποιες επιτυχίες αυτή την περίοδο. Το πρόγραμμα, τα προγράμματα με κεντρική διαχείριση έχουν ε, αυξημένο προπολογισμό. Τα προγράμματα με κοινή διαχείριση ε, ε, έχουν μειωμένο προπολογισμό. Αυτή είναι η τάση. Ε, αυτή είναι μια τάση σε, όλο το, σε όλη τη δέσμη μέτρων. Αυτό διότι η κεντρική διαχείριση είναι κάτι εύκολο, πιο εύκολο να το διαχειριστεί κανείς, είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί, είναι πιο εύκολο να πετύχει αποτελέσματα και γρήγορα και στις περισσότερες περιπτώσεις των προγραμμάτων τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα τα οποία στηρίζονται εύκολα από τις τράπεζες, από τους ιδιωτικούς επενδυτές και το καθεξής. Όλα τα υπόλοιπα αυτά που συζητούμε συνήθως εδώ όταν αναφερόμαστε στην πολιτική συνοχής δεν είναι προγράμματα που μπορούν να περάσουν από τις τράπεζες. Το να συγκρίνουμε προγράμματα όταν τα προτείνουμε ε, αυτό είναι κάτι που να το αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι που αφορά τη διαδικασία. Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργεί η διαδικασία στο μέλλον. Αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης. Έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως, έχουμε τις θέσεις των σκιωδών ε, εισηγητών. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε εκπρόσωπο της Γενικής Δευθύνσεως ΕΚΦΙΝ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον συγητή για την, το σχέδιο γνωμοδότησης όσους συνέβαλαν στη συζήτηση. Πρέπει να, πιστώ, να πείσω πολλούς στην αίθουσα από ό,τι φαίνεται. Θα ξεκινήσω όμως από κάποιες εξηγήσει σχετικά με το στόχο που έχουμε θέσει. Όπως τονίσατε σωστά, Πρόεδρε, αυτό το τμήμα των 100 μελών εκτελείται επιθελοντική βάση. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θελοντικά δίνουν τα χρήματα προς το InvestEU. Ακούσαμε πολλά να αναφέρονται για αποφάσει τοπικής αυτοδιοίκηση, ελεύθερε απόφαση τοπικής αυτοδιοίκηση. Ας αποφασίσουν. Στόχος είναι η διευκόλυνση των συνεργειών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των διαφόρων διαχειριστικών μέσων στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως για προγράμματα στις διάφορες περιφέρειες. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αν κάποια περιφέρεια θέλει να χρησιμοποιήσει το κομμάτι των κρατών μελών το οικονομικό, το κράτος μέλος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τους πόρους της περιφέρειας Δηλαδή δεν είναι ότι η Καλαβρία συμβάλλει στο τμήμα της, ε, Ευρω... Ε, του κράτους και το κράτος χρηματοδοτεί το παιδεμόντιο. Αυτή δεν είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ωφεληθούν τα κράτη-μέλη από αυξημένο όγκο στηριζόμενης χρηματοδότησης. Λοιπόν, έχουμε και κανόνες ακούσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού να αναφέρεται. Πράγματι είναι πρόβλημα και γι' αυτό προσπαθούμε να διαθέσουμε 14 διαφορετικά μέσα με διάφορα κριτήρια επιλεξιμότητας και όλα αυτά να μπουν υπό μια κοινή αιγίδα. Πιστεύουμε ότι συνδυασμό των πόρων μεταξύ του τμήματο των κρατών μελών και του τμήματο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό και οποιαδήποτε ποσό του κάτω μέλου που διατίθεται μέσω του InvestEU θα διατίθεται σε αυτό το κράτο μέλο και το κράτο μέλο αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει στην περιφέρεια που θέλει. Η συμφωνία συνεισφορά μεταξύ κράτου μέλου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια συμφωνία για διάθεση κάποιου στόχου. Δεν θα πηγαίνουν από μια περιφέρεια σε άλλη τα χρήματα. Και θα μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι της DG Regio γι' αυτό. Όταν γίνει η μεταφορά προς το InvestEU, η εκτέλεση στο τμήμα του κράτους μέλους θα ακολουθεί τους κανόνες του InvestEU και θα υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση και έλεγχος. Σύμφωνα με τους δικούς μας κανόνες για το InvestEU και θα υπάρχει και, πιο, και απλούστευση των κανόνων για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Επίσης υπάρχουν και κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα σήμερα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. και τα πιστοτικά μέσα με τις χορηγίες πρέπει να συγχωνευτούν. Είναι περίπλοκος ο συνδυασμός όλων αυτών των πόρων. Από κοινή διαχείριση προς κεντρική διαχείριση. Θέλουμε το τμήμα, μέσω του τμήματος του κράτους μέλους να διευκολύνουμε την κατάσταση και τη διοχέτευση των πόρων. Εάν είμαστε πολύ επιτυχείς, τότε θα έχουν και κίνητρο τα κράτη-μέλη να διοχετεύσουν χρήματα. Και κάτι άλλο. Έχει προθεσμίες ο κανονισμός. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα, επιστρέφουν τα χρήματα στο κράτος μέλος. Δεν μπορούν να είναι σε ένα απόθαμα περιμένοντας για μια συμφωνία εγγύησης να υπογραφεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει εταίρο για την υλοποίηση, εφαρμοστικό εταίρο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επένδυσης και ο σχετικός όμιλος είναι ο εταίρος μας τώρα. Θα επεκταθεί ο αριθμός των φορέων που έχουν πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στις εγγύησεις μας και αυτός είναι ένας υγιής τρόπος ανταγωνισμού η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να επιλέξει τον εταίρο υλοποίηση Και άλλη πρόταση που τα, τα κράτη-μέλη θα υπογράψουν μια συμφωνία συνδρο, συμβολής. Να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Το πρόγραμμά μας είναι ανοιχτό όχι μόνο στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά σε διάφορους τραπεζικούς θεσμούς των κρατών μελών και μεγάλων και μικρών κρατών μελών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εγγύηση. Για μικρά κράτη-μέλη είναι πολύ δύσκολο ε, να έχουμε μεγάλου όγκου προβλήματα που είναι αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη είχε κάνει προσπάθεια να μειώσει τον ελάχιστο αποδεκτό όγκο. Αλλά σε κάποιες χώρες πράγματι αληθεύει υπήρξε πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε τη διαδικασία αξιολόγησης πυλώνα που προβλέπει το δημοσιονομικό κανονισμό ούτω ώστε να βοηθήσουμε τα μικρά κράτη-μέλη και τι διεθνείς τράπεζε που επιθυμούν που μπορούν να έχουν πρόσβαση τον τρόπο στην εγγύηση. να συνεργαστούν καλά με τον όμιλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μπορούν να, είναι, να έχουν σαν διαμεσολαβητή τον όμιλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την περασμένη εβδομάδα οργανώσαμε ένα εργαστήριο πάνω σε αυτό και πολλές χώρες ήταν παρούσες και διάφορες τράπεζες της Κροατίας ήταν παρούσες οι χώρες και ενδιαφέρθηκαν για αυτό το θέμα. Ε, διότι έτσι υπάρχει δυνατότητα αντιμετωπίσεως ε, προγραμμάτων με όγκο που δεν μπορεί να καλυφθεί τώρα. Άκουσα να λέγεται ότι θέλει να γίνει τράπεζα Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε να γίνουμε τράπεζα. Όπως και με το ΕΦΣΥ, Έχουμε διατάξει ό,τι βλέπει έλεγχο και διαχείριση του κινδύνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπολογίζει την παροχή. Αυτό ισχύει και για το ΕΦΣΥ. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο υπολογισμός του κινδύνου και της παροχής δεν βασίζεται σε εισρωή πληροφοριών από έναν εταίρο υλοποίηση, από διάφορους εταίρους που θα έχουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται μία ομάδα προγράμματος που θα εξετάζει κατά πόσο συνεπείς οι πληροφορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητούμε τις πληροφορίες ή την ορθή διαδικασία που ακολουθείται. Είναι με τραπεζική πτυχή που θα εφαρμόζουν οι διάφοροι εταίροι για την ορθή διαχείριση. Εμείς λογοδοτούμε στο Κοινοβούλιο, στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε το χαρτοφυλάκιο που υποβάλλουν οι διάφοροι εταίροι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εξετάζουμε τα, τις υποβολές δεν θέλουμε να καλύψουμε τραπεζικές δραστηριότητε εμείς. Αυτό είναι ήδη απαντήσω στα διάφορα σημεία που ετέθησαν. Κατανοώ τις εκφραστήσεις ανησυχίες. Ελπίζω ότι αυτή η παρέμβασή μου κάπως βοήθησε να διευκρινίσω κάποιες πτυχές και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο της DG Regio, ούτως ώστε να συμπληρώσει τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συμπληρώσω τόσο είπε ο Στη σημερινή συνάντηση ακούσαμε πολλά πράγματα που ακούσαμε και όταν συζητούσαμε το Omnibus. Ε, ακούσαμε λοιπόν προσεκτικά τη συζήτηση και θέλω να εξηγήσω κάποια ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, εδώ μιλάμε για χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν πρόκειται για την επίτευξη ενός πολιτικού στόχου, πρόκειται για την υλοποίηση και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοπιστωτικά μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε προγράμματα και να στηρίξουμε επενδυτικά περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι σε θελοντική βάση γίνεται αυτή η βοήθεια. Δηλαδή οι χώρες μέλη έχουν επιπλέον επιλογές για να χρησιμοποιήσουν ε, ποσά. Όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό βάσει των σημερινών κανόνων, εφόσον θεωρούν ότι είναι σωστή η επιλογή για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Αλλά η κάθε χώρα αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες της. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που αντικατοπτρίζει και άλλες συζητήσεις που έγιναν για το Omnibus είναι ότι δεν πρόκειται για μεταφορά. Άλλο είναι το άρθρο της μεταφοράς. Δεν χάνονται τα χρήματα. Εδώ γίνεται μία συνεισφορά και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η πρόταση της Επιτροπής διασφαλίζει ότι τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο Invest EU παραμένουν στην αρχική πηγή ως δικαιοδοσία. Δηλαδή τα χρήματα έρχονται από ένα πρόγραμμα και πρέπει να φέρουν σε πέρας τους στόχους της περιφερειακής ακριβώς ανάπτυξης τους στόχους της συνοχής. Αν είναι από τη συνοχή, θα πρέπει να συνεισφέρουν στους στόχους της συνοχής. Οι χώρε μέλη διαπραγματεύονται και γίνεται και κατάλληλη αναφορά μετά. Οφέλη υπάρχουν. Η χώρα μέλος αποφασίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο, τη μόχλευση, το ύψος κάλυψης κινδύνου κλπ. Πρέπει να δούνε το ωφέλη κατά περίπτωση. Τέλος, για αυτό που είπατε για τις συνέργειες, την προηγούμενη περίοδο, αλλά και αυτήν, ή το δυνατό να συνεισφέρουμε σε ευρωπαϊκά μέσα. Αλλά είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Αν θέλετε άλλη επιλογή, μπορείτε να το κάνετε με συγκεκριμένους κανόνες και συνεισφέρετε στο Invest EU, αλλά βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, του ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ξέρουμε και από το Omnibus για αυτές τις εξηγήσει. Ήταν χρήσιμο που ακούσαμε την εκθήνη. Παρακαλώ, η συντάκτρια γνωμοδότηση, κυρία Βέστφαλ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τρόπο κάπως ανορθόδοξο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν από δύο χρόνια στο βωμό του ΕΦΣΥ δεν θέλω να θυσιάσω την ε, πολιτική συνοχή. Η συζήτηση που έγινε τώρα επιστρέφει, μας επιστρέφει στην ε, προσπάθεια που έκανε η Επιτροπή μας όλα αυτά τα χρόνια για να απλουστευτούν, απλουστευτούν οι καταστάσεις και να μεταφερθούν στις περιφέρειες στους απλούς πολίτες την απόφαση για το πώς θα ε, δαπανηθούν αυτοί οι πόροι. Δέκα χρόνια είμαι εδώ στην Επιτροπή και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε εργαστεί ευελιξία, απλούστευση και τώρα με τον νέο γενικό κανονισμό και με όλα που σχετίζονται με αυτό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και το είπα από την αρχή. Η δουλειά μου είναι μέσω της γνωμοδότησης να μην θυγεί η διαθροτική πολιτική να διατηρηθεί. Διότι η διαθροτική πολιτική πρέπει να έχει τους επαρκείς πόρους για τις υποδομές, την κλιματική αλλαγή, να δημιουργηθεί εργασία, να στηριχθούν ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια. Δηλαδή πράγματα που είναι πολύ κοντά στους πολίτες. Αυτό είναι κάτι για το οποίο διαμαρτύρεται η Επιτροπή μας. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες, να υπάρχει ορατότητα. Περί αυτού πρόκειται και το ξαναλέω. Θα πρέπει η ζήτηση να συνεχιστεί και να είμαστε ακόμη πιο κατηγορηματικοί και για το Γενικό Κανονισμό θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο. Η Επιτροπή δική μας να έχει πρώτα απ' όλα το Γενικό Κανονισμό και όλες οι άλλες γνωμοδοτήσεις οι εκθέσεις για τους επιμέρους κανονισμούς να ε, συντονίζονται με αυτό. Με την αντιμετώπιση μας για το γενικό κανονισμό. Δεν είναι δυνατόν μια γνωμοδότηση να έχει εντελώ άλλη κατεύθυνση από την ε, άποψή μας για το γενικό κανονισμό. Γι' αυτό όλοι συνεργαζόμεθα εδώ σε αυτή την Επιτροπή για να υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση και είμαι πεπισμένη ότι δεν είναι τελευταία φορά που θα κάνω αυτή τη συζήτηση για την γνωμοδότησή μου δηλαδή αλλά θα τη συνεχίσουμε διότι πρέπει να είμαστε παρκώς κατηγορηματικοί και να τονίσουμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την περιφερειακή πολιτική και θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Οίκον και Μπούτζι είναι οι επί της αρμόδιες. Θα ψηφίσουν τις εκθέσεις τους 19 και 20 Νοεμβρίου. Άρα εμείς πρέπει να ψηφίσουμε επί της γνωμοδοτήσεώς μας στις 25 Οκτωβρίου στην ε, ε, έκτακτη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. Οπότε προθεσμία για τροπολογίες 5η 4 Οκτωβρίου. Αλλά 12 το μεσημέρι. Σας δίνω μισή μέρα παραπάνω. 5η 4 12 το μεσημέρι. Και παρακαλώ να είναι στα αγγλικά οι τροπολογια σας. Αν γίνεται, αν γίνεται. Επαναλαμβάνω. 4 δεκάτου. 4. 12 το μεσημέρι. Και αν γίνεται, αγγλιστή. Θα μας διευκολύνει. Και το τελευταίο σημερινό θέμα, συγγνώμη που έχουμε καθυστερήσει, ανταλλαγή απόψεων επί της προτάσεως Επιτροπής για ένα μηχανισμό για την επίλυση νομικών και ε, διοικητικών προβλημάτων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Είμαστε υπεύθυνοι επί της ουσίας και ο εισηγητής μας ο κύριος Φαν Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στο Ολλανδικά, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γι' αυτό και θα μιλήσω στη μητρική μου, για να μπορώ να διατυπώσω καλύτερα τη σκέψη μου. Λοιπόν, Ολλανδικά συνεχίζει ο μιλητής. Είναι γνωστό σε όλους και όλοι καταλαβαίνουν ότι η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για όλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά είναι ένα διασυνοριακό κομμάτι. Εκεί ζουν πάρα πολλοί πολίτες μας και είναι υπεύθυνο για το 30% του ΕΠ. Το έχουμε δει στην ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θέλει να ενισχύσει λοιπόν την διασυνοριακή συνεργασία. Και όντω υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε αυτήν την συνεργασία. Οι κάτοικοι των διασυνοριακών περιοχών βρίσκονται αντιμέτωποι πάρα πολύ συχνά με εμπόδια. Και στην Ολλανδία το έχουμε αυτό με την Γερμανία ε, που κάτι θέλει η Γερμανία, κάποιο έργο που πρέπει να γίνει και στην Ολλανδία, αλλά δεν μπορεί. Γι' αυτό θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση για τις διασυνορικές αυτές περιοχές, να μπορεί να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και στα έργα χωρίς διοικητικά εμπόδια. Να μην υπάρχουν λοιπόν πια αυτά τα εμπόδια. Προτείνει ένα μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σκοπό. Ένα μηχανισμό που θα έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορεί να γίνεται πιο εύκολη παραμεθοριακή συνεργασία. Υπάρχει δυνατότητα με τα Ίντερεκ προγράμματα βέβαια μέχρι τώρα που χρηματοδοτούν πάρα πολλά ε, προγράμματα. Είναι φυσικά οι προθέσεις πάρα πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά έχοντας συζητήσει με πολλούς ανθρώπους διαπιστώνουμε ότι και με τις καλύτερες προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λύνονται τα προβλήματα. Τώρα λοιπόν, σε θελοντική βάση θα μπορούσε να υπάρχει ένας οργανισμός συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών διασυνοριακά. Φυσικά χρειάζεται επικουρικότητα για να ισχύσει. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιούμε ότι χρειάζεται η συνεργασία των χωρών μελών για να μην υπάρχουν πια εμπόδια στην ε, διασυνοριακή συνεργασία. Προτείνεται λοιπόν αυτός ο νέος μηχανισμός σε θελοντική βάση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Σε θελοντική βάση επιμένω αν μία χώρα μέλη δεν ε, θέλει, δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή αυτόν τον μηχανισμό. Οι χώρες μέλη ανάλογα με πρόγραμμα, ανάλογα με το έργο δηλαδή, θα αποφασίζουν. Θα πρέπει να κοιτάει κάθε χώρα μέλος. Ε, όταν ισχύουν οι δικοί τους οι κανόνες, μπορούν να δεχτούν τους κανόνες της γειτονική χώρας για να υλοποιήσουν ένα έργο. Αλλιώ είναι δύσκολο να πετύχουν το στόχο τους. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αυτό, να τονίζουμε τον εθελοντικό χαρακτήρα της πρότασης. Έτσι λύνονται πολλά προβλήματα και με τις χώρες μέλη και εφόσον εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Στο μέλλον θα πρέπει να μπορούμε να λύσουμε και προβλήματα με το μηχανισμό αυτό που δεν έχουμε υπόψη μας ότι προκύπτουν ακόμα, αλλά θα προκύψουν στο μέλλον με την λύση αυτή à la carte, όπως σας είπα. Βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Να μην υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες όσον αφορά τον θελοντικό χαρακτήρα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. πρέπει να στηρίξουν αυτό το μηχανισμό, πρέπει να αποφασίζουν ποια θα είναι η αρχή που θα είναι η υπεύθυνη να επιθωρεί, να διαχειριστεί αυτό το διασυνοριακό έργο. Στις χώρες Μπενελούξ θα μπορούσαν να έχουν ε, τον μηχανισμό Μπενελούξ ή κάποιον άλλον να προτείνουν. Ο μηχανισμός αυτός πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα για να λύνονται τα νομικά και διοικητικά εμπόδια σε διασυνοριακό πλαίσιο, αλλά χρειάζεται και πολιτική βούληση ώστε να πετύχουμε. Συνεργασία επίσης χρειάζεται μεταξύ χωρών μελών, μεταξύ περιφερειών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι θα προσφέρουμε κάτι καλό στους πολίτες που θα το υποδεχτούν θετικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Φανίστερο εκ μέρους του κύριου Βέλερ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Ο κύριος Βέλερ ήταν εισηγητής για τον grouping mechanism. Την προηγούμενη περίοδο το είχαμε αναπτύξει αυτό. Και πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μίλτεμπεργκ το βλέπει το θέμα, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ένας πρόσθετος μηχανισμός. Προσθέτει κάτι καινούριο. Αλλά για να εφαρμοστεί ένα νέο μέσο, μερικές φορές χρειάζονται 4 και 5 χρόνια για να αρχίσει να λειτουργεί δηλαδή. μέχρι να συνηθίσει ο κόσμος τον τρόπο λειτουργίας αυτού του νέου μέσου. Με αυτό το μέσο λοιπόν είναι όντως καινοτόμο, όντως προσφέρει πολλές δυνατότητες. Και πρέπει να δουλέψουμε πάνω στον έλεγχο της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει αυτό το μέσο. Χρειαζόμαστε ένα hearing πιστεύω. Χτες είχαμε ακρόαση του ΕΛΚ για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, Ιντερνετ και τα λοιπά. Και κάποιοι τους ρώτησα, ήρθαν από τις ε, χώρες ΕΖΕΣ και τα και συμφώνησαν ότι το διασυνεργειακό σώμα αναλαμβάνει αρμοδιότητες που παραχωρούν οι χώρες μέλη δεν περιμένουν ε, ένα νέο μηχανισμό κάθε φορά που θέλουν να συνεργαστούν ε, ε, με το Βέλγιο ή με κάποια άλλη χώρα. Πρέπει να ακούσουμε λοιπόν αυτούς τους φορείς. Ίσως έχουν να δώσουν πολύ σημαντικά στοιχεία και βοήθεια. Δεν θα ήθελα να τρέξουμε. Θα ήθελα πρώτα να κάνουμε μια ακρόαση. Ας ακούσουμε όλους τους εμπλεκόμενους που έχουν εμπειρίες σε αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε με το Interreg και τα λοιπά, από διασυνοριακά έργα, να μας φωτίσουν. Γιατί πρέπει να βιαστούμε. Να ακούσουμε προσεκτικά. Και αυτό που λέτε επίσης. Σωστό είναι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κύρια Κρέλα εκ μέρους της κυρίας Μαρκόβα. Ναι, κυρία Μάρκοβα δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα διαβάσω τις παρατηρήσεις της. Ευχαριστώ για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Αγαπητοί ηγητέ και οι συνοριακός μηχανισμό είναι χρήσιμο εργαλείο και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκε τέτοιε για αποτελεσματική χρήση αυτού. Σε αυτή τη φάση έχω διάφορα σχόλια τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όπως γνωρίζετε. έχουμε λάβει τις θέσεις διαφόρων περι... παραμεροθωρίων περιοχών. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι όσον αφορά τη θελοντική πτυχή του μηχανισμού, κατά πόσο θα είναι ελεύθερη επιλογή ή όχι. Η δεμή Υπάρχει γενικά θετική άποψη όσον αφορά το όλο θέμα. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέους πόρους, στόχος του μηχανισμού είναι να διευκολύνει τη συνεργασία παραμοθωρίων περιοχών και να έχουμε θετική αλλαγή για τους πολίτες μας. Το αποτέλεσμα της διασύνδεσης Κύλου και Στρασβούργου ε, μέσω τραμ δείχνει ότι είναι εφικτή αυτή η συνεργασία. Η γέφυρα μεταξύ Σλοβακίας και Ουγγαρίας είναι ένα παράδειγμα, αλλά αυτά τα έργα και προγράμματα ήδη έχουν δρομολογηθεί αλλά ο χρόνος που χρειάζεται να ξεπεραστούν διοικητικά και νομικά εμπόδια ε, ήταν πάρα πολύ ε, μεγάλος. Δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω διαφορών μεταξύ διαδικασιών διοικητικών που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες ευθύνες σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο. Θέλω να έχουμε μειωμένη γραφειοκρατία και να εστιαστούμε επί συγκεκριμένων προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Η μείωση των νομικών φραγμών θα αυξήσει την παροχή καλύτερων ε, ε, υγειονομικών υπηρεσιών, ε, μεταφορές θα βελτιωθούν, οι επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν. Γενικός στόχος θα πρέπει να είναι αρμονική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε καλό συμβιβασμό σχετικά με αυτό και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ECR, ποιος θα μιλήσει. Ορίστε κυρία μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, μιλώ εκ μέρους του κυρίου Πιετρόφσκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πακέτο για την περιφερειακή πολιτική προτείνει ένα νέο μηχανισμό για την απλούστευση και εξυγχρονισμό της υλοποίηση διαφόρων διεθνών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι χρειαζόμαστε ένα νέο εργαλείο ούτω ώστε οι κανόνες ενό κράτου μέλους να εφαρμόζονται και διασυνοριακά βέβαια με την άδεια των αρμοδίων αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα εργαλείο σε κάθε σύνορο ούτω ώστε οι διοικητικοί φραγμοί στις περιοχές αυτές να αρθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα μέσο το οποίο θα εφαρμοστεί για δραστηριότητες στις δεσυνοριακές περιοχές. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα άρθρο το 9.2 Δέλτα όπου εκεί δεν προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το εργαλείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατόπιν αιτήματος διαφόρων μπλεκομένων φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Νομικά πρόσωπα το ζήτησαν αυτό ε, ε, ε, και οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί για διασυνοριακή συνεργασία. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν στην κατάσταση κατά την οποία το εργαλείο αυτό θα χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλη κλίμακα, όχι μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί η κατάσταση όπου οι κανόνες ενός κράτους μέλους θα εφαρμόζονται συστηματικά σε ένα γειτονικό κράτος μέλος. Νομίζω ότι αυτό θα περιπλέξει πολύ την κατάσταση και ίσως να οδηγήσει σε κάποιες νομικές υποχρεώσεις και αν επομισθείς μια νομική υποχρέωση, τότε αυτό ε, έχει σημασία νομική. Όταν υπάρχει ένα διεθνικό τέτοιο πρόγραμμα, ε, καμιά φορά υπάρχει και κάποια παρέκκληση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, όταν εφαρμόζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εντός της παρέκκλησης μπορεί να εφαρμόσεις κανόνες από ένα άλλο κράτος μέλος ή μπορεί να βρει και κάποια διαφορετική λύση. Να υπογράψει μια συμφωνία μεταξύ, να υπογράψει δύο κράτη-μέλη μια συμφωνία και ένα κράτο μέλο μετά δηλώνει ότι για το συγκεκριμένο αυτό έργο το κράτο μέλο αυτό θα εφαρμόσει μια ειδική παρέκκληση ούτω ώστε οι, οι κανόνε τη γειτονική χώρα να μπορούν να εφαρμοστούν. Εξαιρετικά όμω, εξαιρετικέ περιπτώσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία Ίσως οι κανόνες να αλλάζουν ε, κατόπιν πιέσεων διαφόρων λόμπι ενό ισχυρού κράτου μέλου. Στην Πολωνία μπορούσε να δημιουργηθεί η κατάσταση όπου η Γερμανία ίσω να ασκήσει πιέσει για να αλλάξουν κάποιοι κανόνε. Αυτό είναι ανησυχητικό. Και νομίζω ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να μην αποτελεί καλή λύση, ίσως να είναι κάτι με μεγάλη χρονική διάρκεια να είναι πολύ μακροσκελίστη στη διαδικασία και χρονοβόρα και δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι επικοδομητικό για οποιονδήποτε που θέλει να υλοποιήσει διασυνοριακά ένα πρόγραμμα. Έχουμε πόρους του Interreg και αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός των προγραμμάτων του Interreg διότι χρειάζεται κάποιος χρόνος ούτως ώστε να διανυθεί όλο αυτό το μονοπάτι το διοικητικό που απαιτείται και χρειάζεται και χρόνος για να ζητήσει κανείς χρήματα την υλοποίηση των έργων. Κυρία Χέλπ έχει το λόγο. Ο κύριος Χέλπ. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικό θέμα μας απασχολεί σήμερα. Πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Το κάθε κράτος μέλος δημιουργεί όπως έχει το δικαίωμα το δικό του μηχανισμό. Όταν πρέπει να υπάρξουν κάποια κοινά εγχειρήματα αποφασίζεται πώς θα ε, συντονιστούν αυτοί οι μηχανισμοί και αυτό πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και μπορεί να θέσει εν κινδύνο και την ε, υλοποίηση του προγράμματος. Όταν τα προγράμματα αυτά είναι εντός της Ένωσης είναι απλούστερα τα πράγματα γιατί υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των μηχανισμών αυτών ε, και των διατάξεων μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά εάν αυτά τα εγχειρήματα ενέχουν συνεργασία και με τρίτες χώρες, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Εγώ έχω συμμετάσχει σε προγράμματα συνεργασίας με την Μπελαρούς και νομίζω ότι όταν η Επιτροπή υπογράφει διεθνείς ε, συμφωνίες θα πρέπει να ε, προβλέπει δυνατότητα συμμετοχής ε, τρίτων χωρών σε κοινά προγράμματα αλλά θα πρέπει οι διατάξεις ε, σε περιπτώσεις τέτοιας συνεργασίας ε, να υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιων συνεργασιών γιατί αλλιώ θα έχουμε μεγάλες δυσχέρειες γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να υλοποιήσουμε καλές ιδέες ε, το δυναμικό που υπάρχει και μπορεί κάποιοι να λένε εντάξει υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για διαμεθοριακά προγράμματα αλλά στην πράξη είναι τόσο δύσκολη η εφαρμογή τους που αν είσαι από τη διασυνοριακή περιοχή στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία δεν θα μπει στον κόπο. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να διασφαλίσει όλα τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινέ προσπάθειες να αξιοποιούν κοινέ ε, προσπάθειες. Κοινέ, ε, συγγνώμη, διατάξεις. Η κυρία Νταμάτο, σύντομα παρακαλώ. Πολύ συχνά στην Επιτροπή μας συζητάμε για μηχανισμούς που στοχεύουν στην ε, προσέγγιση της πολιτικής συνοχής ε, προς τους πολίτες και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι μηχανισμοί της Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως ε, δίνουν την εντύπωση ότι εργάζονται. είναι μια αξιολόγηση για δύο χρόνια της λειτουργίας ε, των διαμεθοριακών περιοχών και η Κομισιόν λέει ότι οι διαμεθοριακές περιοχές δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο οι άλλες. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια δεν στηρίζονται αρκετά σε διασυνοριακές περιοχές. Πρέπει λοιπόν να επιληθεί συντόμως αυτό το πρόβλημα. Να λοιπόν σε τι πλαίσιο εργαζόμαστε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τέτοιου μηχανισμούς που να επιτρέπουν να χρηματοδοτούνται επαρκώς οι διαμεθοριακές περιοχές. Και δεν θα λυθούν αυτά τα προβλήματα μόνο μέσω των επενδύσεων Interreg. Οι μηχανισμοί που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια στις διασυνοριακές περιοχές είναι αναγκαίοι. Γιατί έτσι θα στηρίξουμε και μερικέ ε, περιφερειακέ ομάδε. Δεν έχουν νομοθετικέ δυνατότητε να ξεπεραστούν τα νομικά προβλήματα στι περιοχέ. Θα πρέπει να πούμε ότι η προσφυγή σε αυτό το μηχανισμό είναι θελοντική φύσεω. Ένα κάτω μέλο μπορεί να αποφασίσει με ένα άλλα ε, όμορα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να άρουν αυτά τα νομικά προβλήματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς αυτού του μέσου σε απαντήσει σε εθνικό επίπεδο ε, σε άτυπη επίσημη συνεργασία με ένα περισσότερα κράτη-μέλη όμορα. Εν αυτή περιπτώση μπορεί να αποφασίσει να μην χρησιμοποιεί το μηχανισμό που δημιουργείται μέσω του κανονισμού. Λοιπόν, ο μηχανισμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέτρα και υποχρέωση και δήλωση εν αναμονή του σχεδίου εκθέσεω του συγητού θα εξετάσουμε το πώς πρέπει να ε, ανατεθούν οι διάφορες ε, ευθύνες συντονισμού μεταξύ κρατών μελών, ο ρόλος συντονισμού που θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νομική προστασία των ανθρώπων εκείνων που διαμένουν σε μια περιοχή διασυνοριακή. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ναταλή Φερσάουντε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ επιγραμματική παρουσίαση της πρώτας επιτροπής να διευκρινίσω ορισμένα θέματα. Έχοντας ακούσει τον εισηγητή και τους κοιόδης. Πρώτον, τονίζω ότι δεν είναι μια βεβαιασμένη πρόταση ούτε κάτι που απλώς μας κατέβηκε. Έχουμε κάνει μια πολυετή συζήτηση και διάλογο με τα κράτη-μέλη και τους φορείς, πολλούς μάλιστα φορείς διαμεθοριακών περιοχών, ήδη λοιπόν από το 2015. Η πρόταση λοιπόν που υποβάλλουμε είναι κάτι που μας ζητήθηκε από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς Βεβαίω, καλοδεχούμενη θα ήταν μια δημόσια ακρόαση, αλλά νομίζω ότι έχουμε λάβει τόσο πολλά αιτήματα ήδη από περιφέρειες, δήμους και άλλους φορείς αυτών των περιοχών. Έχουμε λοιπόν κάνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης. Ο μηχανισμός αυτός συμπληρώνει κατά την προσέγγισή μας άλλα υπάρχοντα εργαλεία της ε, εργαλειοθήκης ε, συνεργασίας. Είναι η οικονομική στήριξη που δίνεται μέσω του Ίντερεγ. προσφέρει αυτό το μέσο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα διαμεθοριακών νομικών φορέων που είναι αναγκαία για αυτή τη συνεργασία. Αλλά οποιοδήποτε όμιλος διαμεθοριακής συνεργασίας ε, υπάγεται σε μία νομική τάξη. Δεν μπορεί λοιπόν να διαλέξει ποια δικαιοδοσία θα ισχύει. Άρα το τρίτο εργαλείο είναι μια διαδικασία, ένας μηχανισμός για το πώς θα επιλύουν τα κράτη-μέλη θέματα που δεν είχαν καν ενδεχομένω προβλέψει όταν ενέκριναν τους εθνικούς κανόνες τους. Ήθελα να το διευκρινίσω. Για τα σχόλια ότι κάποιες ομάδες πίεσης θα πιέσουν για να γίνουν αλλαγές στην νομοθεσία κάποιου κράτους, δεν νομίζω ότι είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος. Ο κανονισμός μας βασίζεται στην ε, χρηματοδότηση και την πρόθεση προγραμμάτων νέων δημοσίων υπηρεσιών ή υποδομών. Γιατί κάποια ομάδα πίεσης να ζητήσει αλλαγή κάποιου νόμου. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Και για τα εξωτερικά σύνορα. Να τονίσω ότι είναι κανονισμός. Εφαρμόζεται μόνο για τα κράτη-μέλη. Έχουμε λάβει κάποια σχόλια ήδη από την Ελβετία ότι πολλοί θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίω, ε, ευχαρίστως. Αλλά για τα εξωτερικά σύνορα που αναφέρθηκαν εδώ από τον σκιώδη εισηγητή δεν νομίζουμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Αφορά μόνο εσωτερικά σύνορα. Κύριος στόχος του μηχανισμού είναι να αρθούν ορισμένα επίμονα προβλήματα που δεν επιτρέπουν στην ε, ενιαία αγορά να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρουσα διευκρίνηση. Είναι η πρώτη για απόψεων. Ο εισηγητής θα υποβάλει το σχέδιο έκθεσης στις 15 Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι. Ωραία. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε ακρόαση. Αλλά ας δώσω το λόγο στον ε, Σκιώδη. Δεν θέλω να απαντήσω κι εγώ σε όλο. Απάντησε η Επιτροπή φυσικά και δεν πρόκειται για τίποτα βιαστικό. Σημειώνω το αίτημα για ακρόαση, αλλά είδαμε με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Γραμματεία, ότι είναι δυνατόν να προλάβουμε. Οπότε η άλλη λύση που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε είναι να οργανώσουμε ακρόαση. Η ομάδα μου δεν θα ονομάζεται ακρόαση της Περιφερειακής Επιτροπής, αλλά της Άλντε. Και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους, ε, κάποιος από το Cambridge, ο οποίος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και να έχουμε εκεί και με την Επιτροπή ανταλλαγή απόψεων. Δεν θέλουμε να επιβραδύνουμε τη διαδικασία βέβαια, γιατί όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι και είναι πολλά τα μέρη που εμπλέκονται ήδη από το 2015. Οπότε έφτασε η ώρα να φέρουμε αποτελέσματα και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Μην χάσουμε πολύ χρόνο γιατί οι άνθρωποι που ζουν σε διασνοριακές περιοχές δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Πρέπει να δράσουμε. Εννοείται ότι θα λάβω υπόψη με όλες τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Όσοι δεν είναι εδώ πια, πρέπει να πω έτσι κι και για αυτούς ότι το θέμα δεν είναι να δυσκολέψουμε τα πράγματα, ούτε να υποχρεώσουμε τίποτα να γίνεται παντού και πάντα. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να υλοποιούνται τέτοια κοινά προγράμματα με νέο τρόπο. Ωραία. Τότε ο συγητής μα θα κοιτάξει για την οργάνωση τη ακρόαση αυτής. Θα ξανασυζητήσουμε και θα ξανασυζητήσουμε έτσι κι όταν θα παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας στην Επιτροπή μας. Την έκθεσή σας μάλλον, την έκθεσή σας. Φανίστε Θα έπρεπε να μπορούν να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές ομάδες, έτσι δεν θα είναι τη ρέγγια ακρόαση, θα είναι πολιτική ομάδα. Ωραία, συνεχίζουμε τη μεσδιάταξη. διάταξη, διάφορα. Δεν βλέπω τίποτα, ελπίζω να μην έχετε τίποτα, λέει ο πρόεδρο. Ωραία, επόμενη συνεδρίασή μα. θα λάβει χώρα στι 8 Οκτωβρίου το απόγευμα και 9 Οκτωβρίου, πρωί και απόγευμα. Και τώρα έχουμε πολύ σύντομα συνεδρίαση των συντονιστών. Έτσι, να είμαστε καλά οργανωμένοι, παρακαλώ. Παρακαλώ, όλοι οι προσκεκλημένοι, οι άλλοι που είναι παρόντες εδώ και δεν έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες στη συνεδρίαση των συντονιστών, να αποχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.